Dear uh, Κυρίες και κύριοι, ας ε, ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΙΝΤΑ για σήμερα. Ε, το πρώτο σημείο για σήμερα είναι το σημείο 16, παρουσίαση δηλαδή από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του κεφαλαίου εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κορέας. σε αυτήν την ε, συμφωνία ε, με την Κορέα. Δηλαδή για πρώτη φορά έχουμε συμπεριλάβει σε ένα τέτοιο είδος συμφωνία στον λόγο κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο μόνιμος ε, συντής μας για αυτό το θέμα, κύριο Σάινφελτ, προετοίμασε μια σχετική έκθεση και η συμβουλευτική ομάδα ανέφερε ότι στην χώρια νομοθεσία της ε, Νοτιού Κορέας υπάρχουν πολύ σοβαρές παραβάσεις της ε, σύμβασης ε, του ΆΕΛΟ. Και ορισμένες από τις σύμβασεις ΆΕΛΟ δεν έχουν κυρωθεί ακόμα από την Κορέα. Οπότε εκφράστηκε με σαφήνεια η αξίωση να αναλυφθεί η δράση σε σχέση με την ε, Νότιο Κορέα, ακριβώς σε σχέση με τα προβλήματα που μόλι τώρα ανέφερα. Η Επιτροπή απέστειλε μια αντιπροσωπεία στην ε, Νότιο Κορέα και έχω μπροστά μου εδώ και ένα άρθρο από μια εφημερίδα της Νότιο Κορέας η οποία αναφέρεται στην λόγω επίσκεψη ε, της οποίας συγχύθηκε Ματλίν Τουνίγκα και την οποία καλωσορίζω σήμερα εδώ. Ε, και υπήρξε ακριβώς η αξίωση του να ξεκινήσουν ουσιαστικές ε, συνομιλίες ε, μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Αλλά ας δώσω τώρα το λόγο στη Ματλέν για να μας ενημερώσει λίγο πιο λεπτομερό σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Καλημέρα, αξιότιμα μελητές συναδελφοί και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα εδώ να σας ε, ε, παρουσιάσω ε, την ενημέρωση από τη μας πλευρά σε ό,τι αφορά την Νότια Κορέα. Έχω μαζί μου και τον Μάγκελ Φρίμπριχ από την νομική μονάδα και τον Κώστα Κανάε από το Γραφείο Γεωγραφικής Κατανομής. Ανακεφαλαιώνοντας καταρχήν να σας πω ότι η διαδικασία την οποία ακολουθούμε για να ασκήσουμε πιέσει στην Νότιο Κορέα σε ό,τι αφορά την κήρυξη του ΕΕ από το 2011, είναι πολύ μακρά. Και όπω είπατε, εδώ εστιάζουμε σε δύο κύρια ζητήματα. Δηλαδή στην κύρωση των ε, κυρίων συμβάσεων ΑΕΛΟ, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα τη ε, ε, συνάθρηση. Επίση, η δεύτερη αξίωση είναι να συμμορφώνεται με τι βασικέ αρχέ τη ΑΕΛΟ, ακόμα και αν δεν έχει κυρώσει όλε τι συμβάσει. Ε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το, την ελευθερία του δικαιώματο συνεταιρίζεστε. Όπω θα γνωρίζετε, ε, ε κατά την, ε, ε, ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε αναφέρει ότι είχε ξεκινήσει μια συνομιλία, αλλά τότε είχε αναφερθεί από τον τότε Πρωθυπουργό ότι θα ε, κινούνταν προς την κατεύθυνση του μηχανισμού επίλυσης διαφορών, ωστόσο με τον Πρωθυπουργό Μουν τώρα ε, βλέπουμε περισσότερη πρόοδο και με την, ε, σε, επιτρο, σε επίπεδο Επιτροπή Εμπορίου και σε επίπεδο Επιτροπής TSD. Παρότι λοιπόν η νέα κυβέρνηση μου ε, ξεκίνησε με περισσότερη βούληση, με περισσότερη όρεξη αυτή την διαδικασία για την κύρωση από τον προηγούμενο Ιούλιο. Έκτοτε, ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημεία, κάποια εμπόδια, γιατί υπήρξαν κάποιες διαφορετικέ απόψει. Και γι' αυτό η Επιτροπή υπέβαλε ε, ένα αίτημα ε, για την ε, έναρξη διαπραγματεύσεων διακυβερνητικών στις 17 Δεκεμβρίου και το εν λόγω αίτημα από την πλευρά της Επιτροπής είναι δημόσια διαθέσιμο. Ε, η προθεσμία που προβλέπεται για τη διαβούλευση είναι τρεις μήνες, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να ίδρυθεί, να, να, να συγκληθεί ένα πάνελ. η Κορέα απάντησε με ταχύτητα και με θετικό τρόπο απέναντι σε αυτό το αίτημα για την ανάληψη διαδικασίας διαβούλευσης. Και αυτό σε συνέχεια και της επίσκεψη που κάναμε πολύ πρόσφατα, τώρα δηλαδή 21 και 22 Ιανουαρίου ε, στη Σεούλ. Εκεί κάναμε μια σειρά από επίσημες αλλά και ανεπίσημες ε, συναντήσεις ε, με ενδιαφερόμενους φορείς, με συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες αλλά και το τριμερές όργανο της Κορέας το οποίο ακριβώς έχει ως στόχο την εξέβρεση λύσεων σε ό,τι αφορά τα εμπορικά ζητήματα. Όπως είπατε και εσείς, ε, Πρόεδρε, ε, προσέλκυσε τον ενδιαφέρον του τύπου και γενικότερα της ε, του ευρωστινού της Κορέας και θεωρούμε ότι πραγματικά υπάρχει αντίκτυπος ε, των προσπαθειών που κάνουμε, γιατί πολλοί νόμιζαν ότι δεν θα καταφέρναμε κάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ίδιε τι διαβουλεύσει, οι οποίε διήρκεσαν μισή ημέρα, ήταν πολύ χρήσιμε σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη κατανόηση τη νομική συμμόρφωση με τη σύμβαση του ΑΕΛΟ ε, και η Κορέα έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά τη. Η κυβέρνησή της ε, δηλαδή κατέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον προκειμένου να κυρώσει τη σύμβαση ΑΕΛΟ και να τροποποιήσει, να προσαρμόσει αντίστοιχα την νομοθεσία της χώρας πέραν από τη συνέχεια που θα δώσουμε μέσω τη ανταλλαγή πληροφοριών με την Κορέα, βρισκόμαστε σε φάση συζήτηση ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα δηλαδή σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε που θα ακολουθήσει η Κορέα και τι διαδικασίε που έχουμε εμεί ξεκινήσει. έχουμε κάποια συγκεκριμένα ορόσημα μπροστά μας. Καταρχήν στις 17 ε, Μαρτίου ολοκληρώνεται η εκπνέη ναι, αυτή η προθεσμία των τριών μηνών για την διαδικασία διαβούλευσης. Από εκεί και μετά, όπως είπαμε, θα είμαστε σε θέση να ζητήσουμε την εγκαθίδρυση ενός πάνελ. Από εκεί και μετά ένα δεύτερο ορόσημο είναι ο Ιούνιος και αυτό γιατί οι, όσοι γνωρίζουν ε, καλύτερα τα πράγματα ε, θεωρούν πως η όθηση αν θέλετε που έχει δοθεί ε, σε αυτή τη διαδικασία για την κύρωση δηλαδή των συμβάσεων ΑΕΛΟ θα μειωθεί καθώς θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος στην Κορέα πλέον. Σε ό,τι αφορά τέλος τον διάλογο και, στο, και με το ε, τρίμερε συμβούλιο και του εκπροσώπου των εργαζομένων και των εργοδοτών, θεωρούμε πως ήταν πολύ χρήσιμες οι πληροφορίε που ανταλλάξαμε. Θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε τον κοινωνικό διάλογο, ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος ε, κοινωνικός, ε, η απαραίτητη κοινωνική συνένεση για την ε, κύρωση των ναι. προφανώς οι συζητήσεις δεν είναι εύκολες. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν διαφορετικές απόψεις από του εργοδότε. Και η δική μα αξιολόγηση είναι ότι οι επόμενε εβδομάδε και οι επόμενοι μήνε θα είναι κέρια σημασία γιατί στο πλαίσιο αυτό θα ξεκινήσει η συζήτηση των προτάσεων ε, στο Κοινοβούλιο. Θα υποβληθούν δηλαδή τα διαφορετικά νομοσχέδια προ έγκριση στο Κοινοβούλιο. Κατά τη δική μα άποψη, η κυβέρνηση τη Κορέα θα πρέπει να ε, παραμείνει αποφασιστική και όπου χρειάζεται να αναλάβει τι απαλέτε πρωτοβουλίε και να κατευθύνει σωστά την όλη διαδικασία. Και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να εστιάσουν στο στόχο του να επιτύχουν ένα σωστό πακέτο αν θέλετε συνένεση. Ε, δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι υπερβολικά φιλόδοξε και οι οργανώσεις οργανώσει και οι εργοδότε θα πρέπει ε, με ε, σειρά του να υποστηρίξουν την κύρωση τη αλόγου. Και δεν θα πρέπει να προσπαθήσουν οι εργοδότες να αντισταθμίσουν, θα θέλετε, αυτήν την διάθεση που έχουν για να υπάρξει κύρωση του αλλού ε, συμπεριλάβουν και άλλα νέα στοιχεία μέσα στη νέα νομοθεσία. Και αναφέρθηκε από δική μας πλευρά ότι θα πρέπει να περάσει το μήνυμα προς τους ε, αρμοδίους ε, συνομιλητές μας από πλευρά της Κορέας ότι θα πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια από δική τους πλευρά προκειμένου να υπάρξει η κύρωση ε, ε, της ΑΕΛΟ. αυτά λοιπόν, βρισκόμαστε στη φάση των διαβουλεύσεων ε, για αυτούς τους επόμενους τρεις μήνες και τα τέλη Μαρτίου όπως είπαμε θα είναι μια σημαντική περίοδος γιατί μέχρι τότε αναμένουμε να έχουμε καταλήξει σε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα και όπως σας είπα θεωρούμε πως ναι τα πράγματα έχουν κινηθεί προς τα μπροστά αλλά ακόμα υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος Σιάνφελ τώρα έχει το λόγο ως μόνος συζητής. E, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο στόχος της σημερινής συνεδρίασης ε, θα έλεγα δεν έχει προηγούμενο. οι διαβουλεύσεις ε, σχετικά με την Κορέα είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνω είναι χωρίς προηγούμενο. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω μόνο, όχι μόνο την ίδια την πολιτική απόφαση αλλά το σύνολο της συμφωνίας στην οποία αναφερθήκατε. Καταρχάς να υπογραμμίσω και αυτή δεν είναι μόνο δική μου γνώμη αλλά είναι η γνώμη οικονομολόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών αλλά και πολλών ειδικών στην Κορέα η συμφωνία αυτή είναι επιτυχής, επιτυχεστάτη. Και δεν θα ήθελα η επιτυχία αυτή να σκιαστεί από τα θέματα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε εδώ σήμερα. Θέματα ναι τα οποία έχουν τη δική του σημασία αλλά ε, δεν είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της συμφωνίας. Γιατί λοιπόν θεωρούμε ότι είναι επιτυχής η συμφωνία αυτή. Βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια σημαντική καινοτομία στην εξωτερική εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, μιλάω για τα κεφάλαια για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης ε, επαναλαμβάνω ότι είναι επιτυχής σε σχέση με τα αποτελέσματα των οικονομικών συναλλαγών ανάμεσα στις δύο πλευρές, προς όφελος και των δύο πλευρών. Να σας υπενθυμίσω ότι οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κορέα αυξήθηκαν κατά 70% κατά τη διάρκεια της περίοδου διαπραγμάτευσης. Οι δε εισαγωγές από την Κορέα αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της ιδίας περίοδου διαπραγμάτευσης κατά 38%. Είχαμε παρομοίως αποτελέσματα και στις ξένες επενδύσεις προς τις δύο χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Κορέα. 34% οι άμεσες επενδύσεις και 46% από την αντίθετη κατεύθυνση. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε να σταθώ εδώ και να υπογραμμίσω αυτή την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη γιατί δεν θα ήταν σωστό να αποσιωπήσουμε αυτή, την, αυτές τις εξελίξεις. Μιλάμε για μια εμπορική συμφωνία η οποία έχει ένα ξεχωριστό ισχυρό κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη. Τίθενται φυσικά τα θέματα τα οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα οποία καλούμεθα να συζητήσουμε. Η επικύρωση των τεσσάρων συμβάσεων από πλευρά της Δημοκρατίας της Κορέας ε, έχει ε, ξεπεράσει τις προθεσμίες που είχαμε δώσει, όπως επίσης ε, για την ελευθερία της πολιτικής συνδικαλιστικής οργανωτικής δράσης των εργαζομένων η υποχρέωση για την δυνατότητα ύπαρξης συλλογικών συμβάσεων, διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το σύνολο του δημοκρατικού κόσμου και φυσικά τον ελεύθερο αυτό δημοκρατικό κόσμο μπορούμε να πούμε ότι εκπροσωπούμε σε ένα μεγάλο βαθμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό θα θέλαμε η Νότια Κορέα να αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις οι οποίες ε, είναι για μας πάρα πολύ σημαντικές και θα ήθελα η Κορέα να υιοθετήσει τάχιστα τις τέσσερις αυτές συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και ταυτόχρονα όχι μόνο να τις υιοθετήσει αλλά και να τις εφαρμόσει πιστά. Από την άλλη θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η λειτουργία μιας βιομηχανίας στο εσωτερικό ενός κράτους δικαίου και οι κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνουν τις συνθήκες εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, ε, όλη αυτή η ιστορία ανάμεσα στους δύο συμβαλωμένους διαφέρει εμείς έχουμε περάσει από την Ευρώπη κάποιες αλλαγές οι οποίες μας φαίνονται σήμερα προφανείς. Αλλά σε άλλες πλευρές του κόσμου τα πράγματα τα βλέπουν με διαφορετικό μάτι. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτές οι διαφορετικές αξίες, αυτές οι διαφορετικές αντιλήψεις απαιτούν μια εξελικτική διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουν να σεβαστούν τα χαρακτηριστικά της κάθε πλευράς. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μην αναφερθώ μόνο στην οικονομική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και την πολιτική κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται οι πολιτικές σχέσεις έχουν αρχίσει και αλλάζουν. Οι θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αλλάξει άρδεν. Βλέπουμε την εμφάνιση επίσης στη διεθνή σκηνή της Κίνας με ισχυρό τρόπο. Αυτά τα χαρακτηριστικά εν πολλής εξασθενούν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πάρα πολλές, ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Συνεπώς λοιπόν προσπαθούμε να αναλάβουμε δράση, προσπαθούμε να πείσουμε άλλες κυβερνήσεις, άλλες χώρες, έτσι ώστε να συμφωνήσουν μαζί μας και να συμφωνήσουν με τις αντιλήψεις μας. επόμενη λοιπόν για να μην μακρηγορώ. Η συμφωνία αυτή χαρακτηρίζεται σαν μία επιτυχία. Έχει πάρα πολλά και θετικά στοιχεία. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα σημεία τα οποία περιλαμβάνει το άρθρο 13. Ας ακούσουμε τώρα τους ε, σκιώδεις, ο κύριος ε, Σούστε. παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Ε, φοβούμαι ότι εγώ διαφωνώ πλήρως με τον κύριο ε, Σάινφελτ. Ε, ναι, μιλούμε για οικονομική ανάπτυξη, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει η καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Περί αυτού πρόκειται. Εδώ μιλούμε για συνδικαλιστικές οργανώσεις, ε, κρατουμένους Δηλαδή έχουμε ε, φαινόμενα τα οποία είναι εξαιρετικά δυσάρεστα και εξαιρετικά ανησυχητικά. Εδώ στο Κοινοβούλιο μιλούμε για ε, ε, εμπόριο επί τη βάση ισότιμων αξιών και δίκαιων αξιών και λέμε ότι είναι επιτυχής η συμφωνία, όμως έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Θα πρέπει όλα τα τμήματα μιας συμφωνίας να πληρούνται. Το ίδιο ε, λέμε για παράδειγμα και στη Γερμανία και στην Πολωνία και αλλού. Δεν λέμε δηλαδή ότι ε, αν το 80% μόνο της νομοθεσίας πληρείται πρόκειται για επιτυχία ή τηρείται το 100% της νομοθεσίας ή όχι. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για επιτυχία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς την Επιτροπή. Καταρχήν να πω ότι ε, έστω και αυτό τον οδύναμο μηχανισμό, το γεγονός ότι τον, θέσουμε, τον έχουμε θέσει πλέον σε λειτουργία, καλό είναι. Αλλά γιατί το κάνουμε τώρα γιατί αφού δηλαδή γνωρίζαμε από ευθύ εξ αρχή ε, αυτέ τι παραβιάσει οι οποίε υπήρχαν. Γιατί επανειλημμένα έχουμε ακούσει αυτή τη δήλωση ότι δηλαδή η κυβέρνηση της Νότιο Κορέας ε, έχει ξεκινήσει ε, κάποια σκέψη σε ό,τι αφορά την ε, κύρωση. Αλλά δεν βλέπουμε δηλαδή να γίνεται καμία πράξη στην πραγματικότητα. Δεν για παράδειγμα απελευθερώνονται κάποια από τα μέλη που βρίσκονται υποκράτηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Και από εκεί και μετά να σας ρωτήσω, πραγματικά πιστεύετε ότι θα ε, υπάρξει επιτυχής έκβαση αυτής της διαδικασίας, γιατί μόλις τώρα είπατε οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν θα πρέπει να έχουν υπερβολικά φιλόδοξες προσδοκίες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι θα υπογράψουμε ένα χαρτί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής από κοινού με την Κορέα χωρίς να απελευθερωθούν αυτά τα ε, μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Και μετά τι μας είπατε, ότι έχουμε προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο, γιατί από τον Ιούνιο και μετά ξεκινάει μια προκληπλοϊκή ε, περίοδος στην Κορέα. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν υπάρχει δηλαδή καμία ε, ελπίδα από εκεί και μετά να προωθήσουμε τη διαδικασία και γι' αυτό θα πρέπει να αναμείνουμε την επόμενη κορεατική κυβέρνηση για να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε. Και αν είναι έτσι τα πράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριο Σταρμπάτη για το ECR. Εγώ Είμαι, έχω τελείω διαφορετική άποψη από τον κύριο Σούστερ, ο οποίος ε, είπε ότι έχει πολύ διαφορετική άποψη από τον α, α, κύριο Στάινφελτ. Ε, δεν κάνουμε μια ζωή λόγω για ανθρώπινα δικαιώματα και για κοινωνικά πρότυπα τα οποία έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διαδικασία της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι μια διαδικασία μακρόχρονη και το βλέπετε αυτό. Ε, δηλαδή πρόκειται για κάτι το οποίο προέρχεται ε, και συνοδεύεται από την οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή ε, πρέπει να υπάρξει επιτυχία, μπορεί, πρέπει να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη για να υπάρξει και ε, η κατάλληλη εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά πρότυπα. Και σας παρακαλώ, με διακόπτετε κύριε Αφήστε με να πω αυτό που θέλω και συνέχεια μπορείτε να ξαναπάρετε το λόγο. Άρα λοιπόν ε, το βασικό εδώ που θα πρέπει να επιτύχουμε είναι μια καλύτερη κατάσταση. Και πάλι ισχύει εδώ η αρχή τη επικορικότητα. Όταν λοιπόν βρίσκεται κάπω εκεί επί τόπου, μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα τα πράγματα από ό,τι εμεί εδώ στην ε, Ευρώπη. Όμω, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι πάντοτε οι Ευρωπαίοι ε, είναι αρκετά αλαζονικοί Δηλαδή, ε, σε πλαίσιο όλων αυτών των δημιουργών συμφωνιών, ε, πάντοτε θεωρούν πως τα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι καλύτερα, είναι υψηλότερα και θα πρέπει να επιβληθούν. Αλλά είναι διαφορετικές οι ιστορικές διαδικασίες που ισχύουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ε, ε, ερχόμαστε εμείς και θα πρέπει να εφαρμόσετε και να σεβαστείτε τα δικά μας ε, πρότυπα. Δηλαδή αυτό είναι ένα είδος οικονομικού υπεριαλισμού. με αποτέλεσμα οι εν λόγω χώρες ενδεχομένως να στραφούν σε άλλους Δεν μπορούμε δηλαδή, για να το πω ομά, να επιβαλόμαστε απλώ και μόνο επειδή είμαστε ισχυρό εμπορικό εταίρο. Και το είδαμε και σε σχέση με την Ελβετία. Πραγματικά πρόκειται για οικονομικό υπεριαλισμό. Και ε, έτσι κι αλλιώς σε διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ακριβώς ένα και ένα ε, σημείο αναφορά αν θέλετε γιατί ο Τραμπ με την κυβέρνησή του ε, ε, δεν είναι αξιόπιστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο ο σταθερό αν θέλετε σημείο αναφορά, αλλά δεν μπορεί να λέει στους υπολείπους ότι θα πρέπει να εφαρμόσετε τα όσα εμείς εφαρμόζουμε στο δικό μας εργασιακό δίκαιο γιατί πρόκειται για τη μόνη σωστή λύση. Γιατί αν το κάνουμε τότε οι εν λόγω χώρες ενδέχεται να στραφούν σε άλλους, για παράδειγμα στην Κίνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή όπως κάνατε εσείς κύριε Σούστερ συναισθηματικό αν θέλετε χαρακτήρα ε, δηλώσεις. Δηλαδή δεν νομίζω πως είναι σωστή προσέγγιση να λέμε απέναντι στην Κορέα μόνο εμείς έχουμε δίκιο και κανένας άλλος δεν έχει δίκιο. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος Κάρολιν. Ε, εγώ από την πλευρά μου θα συνταχθώ με τον κύριο Σούστερ. Ε, διαφωνώ μαζί σας. Ε, δηλαδή από τη μία πλευρά η Νότιος Κορέα ναι είναι οικονομικά επιτυχημένη αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε και το τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην Νότιο Κορέα και ως ε, σοσιαλίστρα εγώ λέω ότι ναι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους ε. και λέμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε το δίκαιο εμπόριο και ότι το ελόγω εμπόριο δεν είναι δίκαιο το βλέπουμε στην Κορέα. Τι ε, θα σημάνει αυτό τώρα για τις μελλοντικέ μας εμπορικές συμφωνίες. Δεν θα πρέπει να ε, συμφωνούμε σε ό,τι αφορά την κύρωση των βασικών συμφάσεων του ILO πρωτού προβούμε στη σύναψη μια εμπορική συμφωνία. Νομίζω πω αυτή θα ήταν η σωστή άγουσα, ώστε να αποφύγουμε προβλήματα όπω αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και μετά αυτό που ακούμε είναι ότι δεν υπάρχουν κυρώσει οι οποίε θα επιβληθούν. Γιατί νομίζω πω η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή τη κανένα μηχανισμό αποτελεσματικό για να τι επιβάλλει. Άρα θεωρώ πω θα πρέπει να υπάρξει ένα μηχανισμό ο οποίο θα είναι δυνατόν να εφαρμόζεται, ο οποίο θα επιβάλλει κυρώσει και ο οποίο με αυτόν τον τρόπο θα ε, ε, βοηθήσει στην πλήρωση των σχετικών κενών. Ε, και νομίζω πω θα πρέπει να υπάρξει αυτό ο μηχανισμό. Οπότε θα πρέπει, ε, επαναλαμβάνω, να. Ε, εντάξει, εδώ να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε λόγο εμπορική συμφωνία, αλλά στι μελλοντικέ θα πρέπει εκ των προτέρων να συμφωνούμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να υπάρχει ε, ε κύρωση των συμβασιών. Αλλά και από εκεί και μετά θα πρέπει να εξετάζουμε το ποιοι είναι εταίροι του οποίου επιθυμούμε. Είπατε κι εσεί ότι είμαστε ένα ισχυρό εμπορικό εταίρο και γι' αυτόν τον λόγο μπορούμε πραγματικά να ασκήσουμε πιέσει στου υπόλοιπου εταίρου και να λέμε ότι μόνο υπό του εξή όρου επιθυμούμε μια εμπορική συμφωνία μαζί σα και όχι υπό άλλου όχι σε άλλη περίπτωση. Ο κύριο Ρίμπιχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το γεγονός ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς ε, ε, την πρώτη φάση αυτή τη διαδικασία, ε, πράγμα το οποίο βέβαια θα ε, ωφελήσει κυρίως τους εργαζόμενου. Γιατί βέβαια αν υπάρχουν περισσότερε εξαγωγέ προ την Νότιο Κορέα ή μάλλον περισσότερες εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι στη Νότιο Κορέα και έτσι βελτιώνεται η αγοραστική δύναμη, υπάρχουν πιο φτηνά αγαθά στην αγορά και ούτω καθεξής. Άρα νομίζω πως με αυτή τη συμφωνία επιτυχάνουμε η υψηλότερη αγοραστική δύναμη μέσω ακριβώ ε, τη μεταμέση υψηλότερων ε, μισθών. Οπότε νομίζω πω εδώ υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα, όταν οι σοσιαλιστέ. Ε, η σοσιαλιστική ομάδα μα λέει δεν χρειάζεται να υπάρξει μια αναδιανομή, μπορούμε να παραμείνουμε μέσα στην ένδια. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω κάτι τέτοιο, είναι παράλογο. Δηλαδή, τι να την κάνουμε τη συνδικαλιστική οργάνωση αν δεν υπάρχει παραγωγή, αν δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Προσπαθώ λοιπόν να είμαι λίγο πιο ρεαλιστή. Το ζητούμενο εδώ είναι να αναγνωρίσουμε την επιτυχία αυτής της διαδικασίας. Ε, και θα πρέπει βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από μια τέτοια συμφωνία. Αλλά αποτελεί βέβαια και ευθύνη των ε, κοινωνικών εταίρων στα, διάφορε στις διάφορες χώρες. Βλέπουμε δηλαδή ε, το πώς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τιμωρούν τους καταναλωτές οι οποίες για παράδειγμα ανακοινώνουν μία απεργία για παράδειγμα μόνο 24 ε, ε, ώρες πριν ξεκινήσει και το είδαμε αυτό στις ε, αεροπορικές εταιρείες όπου δηλαδή ανακοινώνεται μια τέτοια ευνηδιαστική απεργία και βρίσκονται όλες εκείνες οι οικογένειες οι οποίες ήθελαν να πάνε τις διακοπές τους και απλά περιμένουν στο αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέπουμε οι καταναλωτές να υπονομεύονται με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριο Σόλτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσω και εγώ την ε, Μάντλεν ε, που παρευρίσκεται σήμερα ενώ για να μας ε, ενημερώσει σχετικά με τις διαφουλεύσεις, ακόμα και αν αυτές ξεκίνησαν καθυστερημένα. Μα όμως είναι σημαντικό που ασχολούμαστε με αυτήν την, τις υποχρεώσεις δηλαδή που θα απορρέουν από τη σύναψη μιας τέτοιας εμπορικής συμφωνίας. Και νομίζω που κάποιοι συνάδελφοι θα έμεναν έπληκτοι με τα όσα ακούστηκα σήμερα στην αίθουσα. Δηλαδή υπάρχουν δικαιώματα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία θα πρέπει να σεβόμαστε. Και ναι, μέσα σε αυτά τα δικαιώματα συγκαταλέγεται το δικαίωμα απεργίας. Εάν για παράδειγμα το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια λαμβάνει εξευτελιστικούς μισθούς, μισθούς ε, από τους οποίους δεν μπορούν να επιβιώσουν, τότε έχουν το δικαίωμα να απεργήσουν. Ποιο λοιπόν εργάζεται για 50 ε, ευρώ και 90 σέντι, για 6 ευρώ και 90 σέντι. Άρα λοιπόν εκείνο που τίθεται ως ζήτημα είναι θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι η σχέση των μισθών σε σχέση με την ε, παραγωγικότητα. Και αυτή την πτυχή προσπαθούμε να, να λάβουμε υπόψη μας αυτή τη συμφωνία. Όταν λέμε λοιπόν ότι αυτό το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης και του εμπορίου το συμπεριλαμβάνουμε σε μια τέτοια συμφωνία είναι κάτι που το κάνουμε συνειδητά, γιατί εμένουμε στο, ε, στο δίκαιο εμπόριο για όλους και λέμε ότι θέλουμε να έχουμε μια τέτοια εμπορική πολιτική την οποία εφαρμόζουμε εναντί όλων. Κατά τη συνέπεια θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σωστό το γεγονό ότι η Επιτροπή έναντι των εταίρων μα από την Νότια Κορέα επιμένει στην εφαρμογή αυτού του κεφαλαίου. Και εμείς από δική μας ε, πλευρά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και με τους συναδέλφους μας από το Κορεατικό Κοινοβούλιο προκειμένου να ε, εφαρμοστούν αυτές οι συμφωνίες ε, και το πώς δηλαδή μπορεί η εκτελεστική εξουσία εδώ να παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση και την κύρωση αυτών των συμφωνίων. Νομίζω πως ε, αυτά είναι τα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσουμε. Τώρα, οι ιστορικές και οι πολιτισμικές διαφορές ναι, θα πρέπει να ε, γίνουν σεβαστές και σε, σχέση με αυτό συμφωνώ μαζί σας. Αλλά αυτό βέβαια αφορά του πάντε. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε επειδή μας συμφέρει, ε, επειδή για παράδειγμα η Κορέα ε, έχει ένα παρόμοιο οικονομικό μοντέλο με εμά, οπότε είμαστε λίγο πιο ε, διαλλακτικοί. Ενώ για παράδειγμα, όταν συνάπτουμε συμβάσει με άλλε χώρε, γινόμαστε πιο αυστηροί. Όχι, θα πρέπει να έχουμε την ίδια ε, πολιτική απέναντι σε όλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια επαναλαμβανόμενη συζήτηση αυτή που έχουμε εδώ. Εγώ είμαι απολύτω υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων των ανθρωπίνων και των εργαζομένων αλλά είναι αρκετά δύσκολο, ίσως αδύνατο να δούμε ποια τρίτη χώρα σέβεται τέτοιου είδους πρότυπα αντίστοιχα με τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως ο Καναδάς και άλλες μια-δυο χώρες. Δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με καμία χώρα στον κόσμο αν εμέναμε σε αυτό. εάν δεν συνάψουμε μια εμπορική συμφωνία, αυτό θα είναι δεν θα είναι προς το συμφέρον του συνόλου των εργαζομένων των χωρών αυτών συμπεριλαμβανομένης της Κορέας. Πρέπει να δούμε πού βρισκόμασταν και πού προσπαθούμε να πάμε. Αυτές οι συμφωνίες είναι χρήσιμες για να βελτιώσουμε τις συνθήκες των εργαζομένων και τα δικαιώματά τους, αλλά αν φανούμε υπερβολικά αυστηροί ε, τότε απλώ ε, θα μπλοκάραμε ε, τη δυνατότητά μα να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Ο κύριο Σούστα και πάλι. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τα όσα είπε και ο κύριο Σταρμπάτη σε ό,τι αφορά την ιστορία και τα σχετικά σχόλια του κυρίου Σόλτς, δεν θα τα σχολιάσω. Το ζητούμενο πάντως δεν είναι αν έχω εγώ δίκιο ή όχι. Το ζητούμενο είναι ότι μία τρίτη χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτουν μία συμφωνία ε, μέρη της οποίας δεν ε, εφαρμόζονται. Δεν έχει να κάνει με το αν εγώ θα ήθελα να περιλαμβάνονται περισσότερα πράγματα μέσα σε αυτή τη συμφωνία ή όχι. Πρόκειται για ένα ε, ζήτημα που τίθεται εδώ ω προ το κατά πόσο παίρνουμε τελικά σοβαρά υπόψη μα ε, το κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης ή όχι. Δεν τίθεται κάτι άλλο προς συζήτηση. Η Κόρεα αλλο προ συζητηση η αυτή τη συμφωνία, όπως συνυπογράψαμε και εμείς αυτή τη συμφωνία στο πλαίσιο της σύναψή τη. Ε, και άρα θα πρέπει να υλοποιείται και από τι δύο πλευρέ. Και δεν μου αρέσει το γεγονό ότι ο κύριο Σταρμπάτη δηλαδή σχετιο, σχετικοποιεί κάθε φορά αυτήν την ε, συζήτηση και ε, δείχνει ότι ουσιαστικά δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του αυτό το ζήτημα. Ο κύριο Σταρπαντή. Κύριε Σούστερ, όταν είχε δημιουργηθεί η ΕΟΚ, η Γαλλία ήταν ο ισχυρότερο οικονομικό εταίρο η Γερμανία η οποία δηλαδή ήταν κατεσταμένη από τον πόλεμο έπρεπε να ανακάμψει και ούτω καθεξής. Και η Γαλλία τότε είχε επιμείνει στην εφαρμογή, στην επιβολή των προτύπων της Γαλλίας ε, στη Γερμανία. Και εκεί χρειάστηκε να, να ασκήσουμε μεγάλες πιέσεις προκειμένου να το αποφύγουμε αυτό γιατί είπαμε ότι ιστορικά έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα και μέσα σε πέντε χρόνια, κύριε Σούστερ, τα σχετικά πρότυπα στη Γερμανία ήταν καλύτερα από τα γαλλικά και μάλιστα οι μισθοί είχαν πλέον καταστεί ψηλότεροι από αυτού στη Γαλλία. Άρα λοιπόν αυτό λέω και ξαναλέω. Αυτά τα πράγματα αποτελούν ε, απόρρια, αν θέλετε, τη οικονομική ιστορική ανάπτυξη. Πρόκειται για μια ολόκληρη διαδικασία την οποία δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε έξωθεν. Οι ίδιε οι χώρε είναι αρμόδιε για αυτέ τι διαδικασίε. Και αυτό που υπόθηκε είναι πολύ σωστό θα πρέπει ναι να παραμείνουμε, να, να, να διατηρήσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με αυτές τις χώρες. Αν αρχίσουμε να είμαστε υπερβολικά ε, περιοριστικοί και τους επιβάλλουμε τους δικούς μας όρους, τότε θα στραφούν στην Κίνα άλλοι. Και εκεί βέβαια ξέρετε ποια είναι τα κοινωνικά πρότυπα. Ο κύριο Σόλτς έχει το λόγο. Κύριε Σταρμπάτη, η Κίνα έχει μία ε, νομοθεσία η οποία λαμβάνει υπόψη της σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με τα σχετικά ε, εργασιακά πρότυπα για παράδειγμα λαμβάνεται υπόψη ε, και το ζήτημα του πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον η αγορά εργασία στην Κίνα. Άρα και η Κίνα λοιπόν εξελίσσεται από την πλευρά τη Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε σύγκρισεις εδώ. Η Γερμανία δηλαδή κατάφερε τα όσα κατάφερε ε, με βάση τον προστατευτισμό. Ότι δηλαδή αμέσως μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε προστατευτισμός, ήταν αποκομμένες οι αγορές. Ισχύει αυτό κύριε Σταρμπάτη. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε μια συμφωνία την οποία έχουμε συνάψει. Δηλαδή, περιλαμβάνει λόγω συμφωνία συγκεκριμένε παραγράφου, συγκεκριμένα κεφάλαια, τα οποία έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και το είπαμε από την αρχή. Δεν τα καταφέραμε να είναι δεσμευτικά αυτά τα στοιχεία παντού, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιμείνουμε στην, ε, στη συμμόρφωση. Θα κλείσουμε τώρα τη συζήτηση, λέει ο Πρόεδρο. Θα ακούσουμε την ε, κυρία Μάντλεν και ίσω και στον κύριο Σεν, Σάινφελντ. Νομίζω ότι μάλλον πλησιάζουμε προ τι εκλογέ Τι λέτε εσείς. Μαντλέν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, έχοντας ακούσει τους ομιλητές, ο καθένας λέει ε, ε, πράγματα ε, που συμπεριλαμβάνουν στοιχεία προς τα οποία συμφωνώ. Κατά την άποψή μας η FTA υπήρξε επιτυχής. Από το 2011 είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν θα έλεγα ότι σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης όλα πάνε άσχημα. Υπάρχουν προβλήματα περιβαλλοντικά, υπάρχουν προβλήματα κοινωνικής υπευθυνότητας, που συμπεριλαμβάνουν και τα εργασιακά ζητήματα, αλλά και εντός του εργασιακού πεδίου έχουμε κάποιες θετικέ εξελίξεις. Η εικόνα δεν είναι τόσο μαύρη και σκοτεινή. Αυτό που είναι κακό ε, είναι ότι μιλούμε ακόμα για επικυρώσει των συμβάσεων ILO από το 2011, δηλαδή χρειάζεται υπομονή. Η Κορέα έχει τη δική της παράδοση και το δικό της σύστημα. Μιλούμε όμως για μια χώρα μέλος του Άσα που είναι ε, υποχρέωσή της να συμμορφούνται προς τις διατάξεις ΑΕΛΟ. Πέραν αυτού, καθότι υπάρχει και η Αμερικανική νομοθεσία για τη δέωση επιμέλεια, ε, γίνεται σχετικός έλεγχος ε, και στην Νότια Κορέα. Τώρα, ακούστηκαν σχόλια για το μηχανισμό μελλοντικών κυρώσεων κτλ. Ε, η άποψή μας είναι γνωστή, δεν είμαστε βέβαιοι ότι αυτό είναι το καλύτερο σύστημα για καλύτερη προσέγγιση. Εν πάση νομίζω ότι στου ερχόμενου μήνες έχουμε μια πολύ καλή δυνατότητα να επιφέρουμε αλλαγή με ένα μηχανισμό που θα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά όχι μόνο ε, σε TSD αλλά είναι κάτι το πρωτόγνωρο για τις ε, συμφωνίες των συναλλαγών, παρότι βεβαίως ε, δεν πρέπει να έχουμε την εντύπωση ότι μια FTA, μια ε, τέτοια συμφωνία θα λύσει τα πάντα. Ας μην είμαστε αφελείς. Και δεν είμαστε. Για τον κύριο Σούστα αμφιβάλλεται για το τι θα κάνουμε το Μάρτιο, μήπω αυτά αξίζουν τον κόπο ή όχι κτλ. Νομίζω ότι το κρίσιμο, η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να δουλέψουμε, είναι αν έχουμε εντοπίσει μια στάση ανάληψης ευθύνης, υπευθυνότητος δηλαδή από πλευράς της τρίτης χώρας. και γνώση άγνοια των υποχρεώσεων εναντιμών και του ILO. Ο κύριος Μουν είπε ότι θέλω να επικυρώσω. Ε, αυτό το θεωρούμε σημαντικό και βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχει μια διαδικασία, μια κίνηση, υπάρχει μια κυβέρνηση που επιθυμεί να τα κάνει αυτά, αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια, αλλά και μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων ε, υπάρχει ενδιαφέρον. Και οι επιχειρήσεις ακόμα αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επικυρωθεί η σύμβαση. Και επομένω, ναι, εμεί πιέζουμε την Κορέα και μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά το πιο σημαντικό και πιο αποτελεσματικό είναι η Κορέα να το κάνει αυτό από μόνη τη. Αυτά ήταν τα κυρίως ε, σχόλια μου. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Ε, θα επανέλθουμε σε ερχόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ κύριος ε, Σάινφελτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, Κοιτάξτε, θα είμαι ειλικρινής πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα, ανοιχτή, ειλικρινής και ευχαριστώ όλους τους παρεμβαίνοντες. Βλέπουμε βέβαια δύο διαμετρικά αντίθετες θέσεις. Και εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ στο μέσον μεταξύ αυτών των άκρων. Ε, ο θεμελιώδη στόχων των συμφωνιών ε, των εμπορικών και των επενδυτικών ε, ακούμε ότι είναι να εξασφαλίσουμε εργασιακή νομοθεσία. Σέβομαι την απόψή σα, αλλά πρέπει να γνωρίζετε το εξή. Δεν υπάρχει κανένα σημείο στη γη, καμία χώρα στη γη, όπου οι άνθρωποι ζουν υπό πιο δεινές συνθήκες εκτός από εκείνες τις χώρες οι οποίες δεν εμπορεύονται με το υπόλοιπο του κόσμου. Ε, εκεί δεν γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου και εκεί έχουμε τα ελάχιστα πρότυπα προστασίας κοινωνικής και εργασιακής. Εμείς έχουμε αναπτύξει μία εμπορική πολιτική, μία εμπορική στρατηγική, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις, στα οικονομικά ζητήματα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες των ε, χωρών αυτών εταίρων και καθόλου δεν λέω βεβαίω ότι η Νότιος Κορέα είναι μία από αυτές τις κλειστές κοινωνίες που δεν εμπορεύονται είναι βεβαίως και ανεπτυγμένη και βεβαίως μια ανοιχτή κοινωνία. Όμως πάντα το νόμισμα έχει δύο όψεις. Έχουμε οικονομικές επιτυχίες που πάντα διαχέονται το trickle down που λέμε για να συνεννοούμεθα. Από την άλλη πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιες από τις προσδοκίες μας δεν έχουν υλοποιηθεί και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ε, πρέπει να συνεχίσουμε μια συζήτηση με την Νότιο Κορέα με θετικό πνεύμα και φιλικά. Σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, Ναι. Είμαι σίγουρο ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, αλλά με αυτό έχουμε ολοκληρώσει με το 16 και θα πάμε στο 17. Ο κύριος Φίζας αντικαθιστά τον κύριο Σαλαφράνκα για κάποιες ε, προϋποθέσεις GATS. Και σας δίνω απευθεία το λόγο. Θα ήθελα να πάρω το λόγο εξ ονόματος του Ινιάσιο Σαλαφράγκα, ο οποίος βρίσκεται στην Νικαράγουα στα πλαίσια μιας ε, αποστολής ε, έρευνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ε, Νικαράγουα και γι' αυτό τον αντικαθιστώ. Είναι τεχνικό το θέμα, κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη σε σχέση με τη Διεθνή Συμφωνία Υπηρεσιών και Αγαθών με συγκεκριμένο περιεχόμενο για κάθε κράτος μέλος που αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1994. Οι ειδικέ διατάξεις τώρα για τρεις χώρες οι οποίες ενετάχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1995 και το 2004 έχουν ήδη γίνει δεχτές και αυτό έχει δημιουργήσει μια περίεργη κατάσταση και μια νομική ανασφάλεια. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια πρόταση απόφασης προς το Συμβούλιο ερχόμενη σε συμφωνία με τα υπόλοιπα μέλη του ΓΚΑΤ έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες έγιναν μέλη το 1995 και το 2004 να ενταχθούν πλήρως στη συμφωνία. Εμείς είχαμε απορρίψει την πρόταση η οποία είχε γίνει το 2007 λόγω έλλειψης διαβούλευσης. Λοιπόν, λόγω πολλών διαδικασιών δύσκολων θα έλεγα, το Συμβούλιο δεν είχε μπορέσει να ολοκληρώσει τα συμπεράσματά του και γι' αυτό χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλήξει σε συμφωνία. Τώρα βέβαια η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη Σιγκαπούρη έχει δημιουργήσει μια νομολογία σε σχέση με το καθεστώς αυτό ιδιαίτερα στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπώς επί τη βάση αυτής της αποφάσεως παρουσίασε μια νέα λύση και ζητείται εδώ η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόταση αυτή ορίζει τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν στα διάφορα κράτη-μέλη και να ενημερωθούν οι λίστες προϊόντων και υπηρεσιών για να προχωρήσουμε σε μια πλήρη τώρα τελική μορφή καταλόγου των αγαθών και υπηρεσιών. Ζητά ο κύριος Αλαφράνκα να εγκρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διασφαλίσουμε την νομική βεβαιότητα και ασφάλεια μιας διαδικασίας η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από το 2004 αλλά ακόμη και από το 1995. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λυθεί το θέμα για τις χώρες που έγιναν μέλη μετά το 2004. Είναι τεχνικό κυρίως το θέμα, αλλά ζητούμε τη σύμφωνη γνώμη. Δεν έχει ζητήσει κανεί το λόγο. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Η παρέμβαση του κυρίου Φίσα εξ ονόματος του κυρίου Σαλαφράγκα έχει νομίζω εξηγήσει σαφώς το τι έχει προηγηθεί του θέματος αυτού το οποίο είναι σε εκκρεμότητα από το 2004. Να επιμείνω στο ότι η κατάσταση έχει δημιουργήσει κάποιες παρενέργειες δυστυχώς οι χώρες οι οποίες έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1995 και το 2004 δεν καλύπτονται ε, πλέον ε, στις ε, συζητήσεις οι οποίες έχουν ακολουθήσει τα ΓΚΑΤ. Αυτό σημαίνει ότι κάποια μεμονωμένα μέλη έχουν αρνηθεί στο να προχωρήσουν στην τελική υιοθέτηση των καταλόγων και αυτό ε, έγινε προφανές όταν προσπαθήσαμε να ολοκληρώσουμε τις συμφωνίες αυτές ε, μετά το 2007. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα και στα πλαίσια του ΠΟΕ που μας α, ε, θεωρεί ανίκανους ουσιαστικά να υιοθετήσουμε μια απόφαση, να εφαρμόσουμε συγγνώμη μια απόφαση η οποία στην ουσία στην αρχή κάλυπτε μόνο 12 από τις 28 σήμερα χώρες. Τώρα λοιπόν και κάτω από τη συνθήκη της Λισαβόνας η υπογραφή, η σύναψη αυτών των συμφωνιών έχει γίνει πλέον αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αναθεωρημένες αποφάσεις από πλευράς του Συμβουλίου έτσι ώστε να επικυρωθούν οι συμφωνίες αυτές που έτσι και αλλιώ έχουν υποστηριχθεί πολιτικά πλήρως από το Συμβούλιο. Να διευκρινίσω ότι οι προτάσεις αυτές είναι ταυτόσιμες περίπου με αυτές τις οποίες είχαμε κάνει το 2007, οι οποίες είχαν γίνει δεκτές από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο η διαφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση η οποία είναι η νομική βάση η οποία έχει διευρυνθεί για να λάβει υπόψη της πλέον και την τελευταία συνθήκη. Ζητάμε λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράσει το ταχύτερο δυνατόν γιατί επαναλαμβάνω ότι η πρότασή μας δεν προσθέτει τίποτα επί της ουσίας, απλά διαδικαστικά μας επιτρέπει να τακτοποιήσουμε την κατάσταση στα πλαίσια των σχέσεων ΓΚΑΤ. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο. Φυσικά ε, θα δράσει το ταχύτερο δυνατόν σε σχέση τουλάχιστον με το ε, Συμβούλιο. Κύριε Φίσας, θέλετε κάτι να πείτε? Όχι. Καλώς, η προθεσμία είναι 25 Ιανουαρίου, 12η μεσημβρινή. 18. ένταξη της Κροατίας στις συμφωνίες με το Μεξικό. Η κυρία Πινέιρο δυστυχώς είναι αδιάθετη και γι' αυτό θα σας διαβάσω τις παρατηρήσεις της. Το πρωτόκολλο αυτό ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ΠΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ένταξη της Κροατίας στην εσωτερική αγορά η έκθεση αυτή είναι τεχνική κατά κάποιο τρόπο, η εισηγήτρια. Θα ήθελε όμως να υπενθυμίσει τα εξής τα οποία έχουν σημασία για το Κοινοβούλιο. Πρώτον, βελτιωμένη ανταλλαγή ενημερώσεων ανάμεσα ε, στα θεσμικά όργανα καθ' όλη τη διάρκεια ε, ισχύω των συμφωνιών. Και αυτό αναφέρεται όχι μόνο για τις μίζωνες ε, λεγόμενες ε, ε, διαπραγματεύσεις, αλλά και τις τεχνικές συμφωνίες. Όλες οι αποφάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται και στη συμφωνία, σαν παράδειγμα απόφαση του Συμβουλίου για τις μπανάνες, για όλα αυτά απαιτείται πλήρης ενημέρωση. Δεύτερον, η πληροφόρηση αυτή, η ενημέρωση αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει μόνο για, την, ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά γενικότερα για τους κοινωνικούς εταίρους, τους εμπλεκομένους και την κοινωνία των πολιτών. Αυτές ε, ε, οι λεπτομέρειες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες επίσης και στο ευρύτερο κοινό. Και αναφερόμαστε κυρίως στην απόφαση που πήρε το Συμβούλιο σχετικά με τις επιπλέον ποσοστώσεις για τις μπανάνες και που δεν είναι βέβαια τμήμα του συγκεκριμένου πρωτοκόλου. Συνεπώς δεν υπόκειται σε έγκριση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τρίτον και τελικά, ο εισηγητής, η εισηγήτρια μάλλον, θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αυτής θα πρέπει να είναι περιορισμένη και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει χωρίς την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις τις οποίες έχει κάνει η συγγήτριά μας. Δεν έχει Α, ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να πω την υποστήριξη από πλευράς μας, από πλευράς της πολιτικής ομάδας, την πρόταση της κυρίας Πινέιρο. Νομίζω ότι επιτρέπεται επιπλέον 2.000 τόνοι για το Μεξικό ε, το οικονομικό αν θέλετε αντίκρισμα δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό μιλάμε για 50.000 ε, τόνους συνολικά ε, εκ των οποίων ένα πολύ μικρό ποσοστό καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία δυνατότητα διαφωνίας με τη συγκεκριμένη πρόταση Καλώς δεν υπάρχει κάποιος άλλος που έχει ζητήσει το λόγο συνεπώς θα ανακοινώσω τώρα την προθεσμία για τις τροπολογίες. Είναι 25η Ιανουαρίου και αυτή κατά τη 12η μεσημβρινή. Τώρα περνάω στο επόμενο θέμα. Είναι το 19. Είναι η αντιπροσωπεία μας στην Χιλή. Η επίσκεψη στη Χιλή έγινε στις 18 μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Ήταν μια αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου, συναντηθήκαμε με 8.000 υπουργού και πάρα πολλού συναδέλφου βουλευτές. Ήταν μια διερευνητική επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον εξυγχρονισμό της εμπορικής συμφωνίας με τη Χιλή. Έχει πράγματι υπάρξει σημαντικότατη πρόοδος οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής έχουν προωθηθεί ε, και θεωρούνται πρότυπο διεθνές. Έχουν εισαχθεί και συμπληρωθεί νέα στοιχεία τα οποία είναι διαφανέστατα. Οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης ήταν επίσης διαφανείς Δημοσιεύθηκαν όλα τα έγγραφα μετά την πρώτη συμφωνία. Υπάρχει επίσης και ένα επιπλέον κεφάλαιο για την ισότητα αμοιβή. Ξέρουμε ότι η Χιλή έχει ένα Υπουργείο Ισότητας των Φύλων και γενικά οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα με υψηλή ταχύτητα. Επί τη βάση λοιπόν της σωστής κατανόησης, της αμοιβαίας κατανόησης με τη Χιλή, Ε, και είναι φυσικά δύο εταίροι οι οποίοι είναι πάντα υπέρ της ε, συνέχισης ε, σε λειτουργία, της λειτουργίας του πολυμερούς διεθνού συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε τους εταίρους να συνεχίσουν την πορεία αυτή βασισμένη στις επιτυχείς διαπραγματεύσεις στο παρελθόν. η εμβάθυνση, εν πάση περιπτώσει, της σχέσης με τη Χιλή είναι ένα υπόδειγμα, όχι μόνο για τη Λατινική Αμερική, αλλά ε, παγκόσμια. Έχουμε και ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον για το λίθιο που παράγεται στη Χιλή και σχετικά με την ε, ηλεκτρονική μορφής ε, κινητικότητα υπάρχει και μια συγκεκριμένη αναφορά στο ειδικό ενδιαφέρον της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει αυτές είναι οι παρατηρήσεις τις οποίες είχα να κάνω και θυμίζω είναι δυστυχώς ασθενής η κυρία Πινέιρο και δεν μπορεί να είναι παρούσα. Τι λέει. Ο κύριος Σάινφελτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, ευχαριστώντας θερμά όλους τους διοργανωτές συμπεριλαμβανομένους της γραμματείας ε, ε, η επίσκεψη ήταν πραγματικά επιτυχέστατη και απολύτως εντός χρονοδιαγράμματος. Ε, πηγαίνοντας τώρα στα θέματα επί της πιστεύω ότι η Χιλή ε, είναι πράγματι μια πολύ σημαντική χώρα για όλους μας, όχι μόνο για τους λόγους που αναφέρατε, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια χώρα ηγέτη ε, σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης στη Νότια Αμερική, προάγει επίσης τις αξίες ε, που μας ενδιαφέρουν, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Και μετά από την ε, οικονομική κρίση η χιλία αναπτύσσεται σε ένα σταθερό 4%. το οποίο αμέσως μάλλον μετά την κρίση ε, κατάφερε να αναπτύσσεται κατά 4 και πλέον κατά 6 με 8% που είναι μια σημαντική οικονομική μεγέθυνση. Είναι ένα πολύ σημαντικό λοιπόν εταίρο. Ως προς την ίδια τη συμφωνία, κατά τη διάρκεια τη συνάντησή μας ε, σε διάφορα επίπεδα, και να υπογραμμίσω εδώ ότι συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους της κυβέρνησης, τον πρόεδρο, με ΜΚΟ, με συνδικαλιστικές ενώσεις, και με ενώσεις ε, διαφόρων εθνικών ομάδων ή στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν ε, σημαντικό ενδιαφέρον από όλους αυτούς τους ενδιαφερομένους ε, για τη συμφωνία. αλλά κάπως απομακρύνονται από το υπερφιλόδοξο ίσως επίπεδο της φιλοδοξίας το υπερβολικά υψηλό επίπεδο της φιλοδοξίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καθώς συζητούσαμε προηγουμένως ε, το θέμα της Νοτιού Κορέας, πρέπει να δούμε αυτό το θέμα της προσδοκίας, των προσδοκιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι με τους οποίους συζητήσαμε μας είπαν ότι η συμφωνία είναι πολύ σημαντική, έχει ε, καταλήξει σε μια πολύ σημαντική οικονομική ανάπτυξη και καλή συνεργασία μεταξύ Χιλής και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φαίνεται ότι τα οικονομικά ζητήματα είναι αυτά που ενδιαφέρουν τους εταίρους, το οποίο ισχύει και για άλλες χώρες ε, στην Νότια Αμερική, αλλά και ε, για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Και βέβαια όλες αυτές οι χώρες διατηρούν οικονομικές και εμπορικές ε, σχέσεις και επαφές και με την Κίνα και αυτό πρέπει να το διατηρούμε υπόψη διαπραγματευόμενοι συμφωνίες πρέπει να μην ξεχνούμε ότι συνολικά το, το πλέγμα των σχέσεων μεταξελίξεται. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, δεν βλέπω ε, κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο. Θα έχουμε ούτως ή άλλως γραπτή έκθεση αρκετά σύντομα. Και μπορούμε να πάμε στο σημείο 20 που είναι η πρώτη ε, ψηφοφορία για σήμερα, πριν ξεκινήσουμε, να κάνουμε μία δοκιμή. Ας δοκιμάσουμε τώρα παρακαλώ. Άρχεται το τεστ. And... <laughs> The test mode is closed. Πέρας της δοκιμαστικής ψηφοφορίας. Ενεκρίθη, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, όλα καλά. Πάμε λοιπόν στο 20, όπου έχουμε τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες 32, 33 και 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ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 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρα 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τι έχουμε τώρα 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να δοκιμάσουμε παρακαλώ, ψηφίστε. Την 106. And the vote is closed. Πέρας. Ναι, εγκρίνεται σαφώς 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ Α, το συγγνώμη, μου διέφυγε. 109 πρώτα. 109 109 λοιπόν. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Χωρίς εμφιβολία. Αποχές λέει τώρα πρόεδρος. «116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται». Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές να δοκιμάσουμε να παρακαλώ την 23 άρχεται η ψηφοφορία And the vote is closed. πέρας ε, ξεκάθαρα απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές. Να δοκιμάσουμε την 1, παρακαλώ. And the vote is closed. And it's adopted. Εγκρίνεται. ε, δύο υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε τη 2 παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η ένα είχε εγκριθεί, έτσι. Η τρία όχι. Άρα πέντε. Υπέρ. Κατά. αποχές Απορρίπτεται. Έξι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και Τελική ψήφος παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και πάμε τώρα στο 21. Το θέμα της συνένεσης. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα και δύο είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται και ηλεκτρονικά πάμε να ψηφίσουμε για το σύνολο παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. και θα πάμε στη δεύτερη έκθεση για τη Σιγκαπούρη, την IPA. Η πρώτη τροπολογία είναι η συμβαστική 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές όχι, α, συγγνώμη λέει ο 34. 34 υπέρ λοιπόν. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 τώρα υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48. Καταπίπτει η πρώτη φράση, αλλά θα ψηφίσουμε για τη δεύτερη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, και πάλι. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά,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 αποχές απορρίπτεται. Δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πέντε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 8 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 9 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 10 υπέρ κατά άποχες Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 10, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεκαοχτώ λοιπόν υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε τώρα επί του συνόλου της ε, πρότασης, της έκθεσης, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στο σημείο 23. Θέλετε να θέσετε κάποιο ζήτημα, συνάδελφα. Ε, πρόεδρε, έκανα λάθος στην τελική ψήφο της προηγούμενης σύμβασης. Αντικαθιστώ ε, έναν συνάδελφο που είναι υπέρ. Αλλά ήθελα απλώς να είναι συνεπής η, στάση που τήρησε. Ο, πρέπει να κοιτάτε τον κατάλογο των ψηφοφοριών, έτσι, και όχι τους συνα... άλλους συναδέλφους. Δεν ψηφίζουμε. Πολύ ωραία. Στο συγγνώμη. Ε, δεν εμφανίστηκαν στη δική μου οθόνη τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Α, εμφανίστηκαν στις οθόνες των υπολείπων. Καλώς, μάλλον ήμουν αφηρημένο. 25 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, καμία εποχή και εδώ είχαμε την δήλωση που έκανε μόλις τώρα ο συνάδελφος για μία ψήφο υπέρ. Βλέπουμε πως ε, ολοκληρώνεται σιγά σιγά η βουλευτική μα θητεία, αυξάνεται η κούραση και ούτω καθεξής. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 23 τη ημερήσια διάταξη. Ε, καταρχήν έχουμε τρεις ε, ταυτόσιμε τροπολογίε, 5, 6 και 7. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τρει ακόμα ταυτόσιμες. 2, 3 και 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, α όχι, η 1 καταπίπτει. Και τώρα ψηφίζουμε επί του συνόλου της πρότασης, άρχεται η ψηφοφορία. Okay, and the vote is... Εγκρίνεται λοιπόν με την ίδια πλειοψηφία όπως στην προηγούμενη, στο προηγούμενο σημείο. Περνάμε στο σημείο 24 λοιπόν. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς. Συμβαστική τροπολογία λοιπόν 1 εδώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε τη συμβαστική 4 για να είμαστε σίγουροι. Άρχεται η ψηφοφορία. ΕΡΑ της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου της πρότασης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν με σαφή πλειοψηφία. Περνάμε στο σημείο 25. Η θέσπιση του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας. Η πρώτη τροπολογία είναι η 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά Α, όχι, 37 υπέρ, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος, κατά τώρα, Αποχέ. Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνουμε μία από κοινού ευσοφορία για τις τροπολογίες 38 έως 44 έχουν υποβληθεί από τον ίδιο συντάκτη. Έτσι. Χάιντι, ρωτάει ο πρόεδρος, συμφωνείς. Ναι, Καλώ. Μαζί με την 37 λοιπόν. 37 έω 44 ψηφίζουμε επί όλων αυτών των τροπολογιών. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Α, όχι. Ζητήθηκε ονομαστική ψηφοφορία για την 54. Παρακαλώ. Vote is απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε, να ελέγξουμε τη 19 λοιπόν ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται. Γι' αυτό σας ζητώ να σηκώνετε ψηλά τα χέρια σας. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάλι ονομαστική ψηφοφορία έχει συντηθεί εδώ για την τροπολογία 20, λέει ο Πρόεδρος, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και μία ακόμα ονομαστική ψηφοφορία. Για την 71 λοιπόν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται και τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά επί του συνόλου, επί του συνόλου της πρότασης άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται λοιπόν με μεγάλη πλειοψηφία τα συγχαρητήριά μας. Περνάμε στο σημείο 26 και την τελευταία ψηφοφορία για σήμερα με ουσιαστικά ένα μόνο σημείο σε ό,τι αφορά μια κατεξοδότηση πράξη. Άρχεται λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της σύστασης. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με συντριπτική πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας παρακαλώ, όποιοι θέλετε να αποχωρήσετε τώρα από την αίθουσα, να το κάνετε σιωπηρά. So, quiet, please, please, quiet. So, next. Σας ευχαριστώ. Our monitor. 27 η έκθεση της Επιτροπής ε, Εποπτείας Παρατήρησης. Δημιουργήσαμε τις ομάδες αυτές για να μπορούμε να συζητάμε σε βάθος τις διαπραγματεύσεις τις οποίες εξελίσσονται και στις οποίες συμμετέχουμε. Οι συζητήσεις σας παρακαλώ εκτός εθούσης. Είχαμε λοιπόν μια συνάντηση της ομάδας για τη Χιλή στις 4 Δεκεμβρίου μιας και είχαμε την έκθεση ε, για την επίσκεψη, δεν χρειάζεται εδώ έκθεση σε βάθος. Έχουμε την ομάδα ε, παρατήρησης των εξελίξεων με την Τινησία στις 8 Ιανουαρίου. Δυστυχώς όμως η κυρία Λαλόντ δεν είναι ανάμεσά μας σήμερα. Είχαμε επίσης και την, ε, την Αυστραλία. Α, Μόζα ε, έφυγε και αυτός από την αίθουσα, δεν παρουσίασε τίποτα. Ήταν μια συνάντηση με τον Αυστραλό Υπουργό Εμπορίου στις 22 Ιανουαρίου. και την ίδια μέρα έγινε μια συνεδρίαση της ομάδας για τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ. Ε, τα ίδια θέματα αυτά τα καλύψαμε χτες με τον κύριο Ντεμαρτή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά ερώτηση ή κάποια παρατήρηση, οπότε αφήνουμε το θέμα αυτό. Πηγαίνουμε τώρα στο 28-29. για την επιλογή των μελών ε, στα Διεθνή Δικαστήρια για τις Επενδύσεις και θα δώσω το λόγο στον ε, ειδικό για, τα, για τις επενδύσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει το λόγο. Καλημέρα σας αγαπητά μέλη, με τη σύμφωνη γνώμη σας θα καλύψω και τις διαδικασίες επιλογής του ICS και το επόμενο θέμα για το πολυμερές δικαστήριο για τις επενδύσεις. Για το πρώτο σημείο, για την διαδικασία επιλογής. Αφορά τις διαδικασίες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή μελών ε, για όλες τις συμφωνίες τις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΣΕΤΑ, ε, Συμφωνία της Σιγκαπούρης. και μελλοντικές συμφωνίες. Στείλαμε κάποια έγγραφα στην Επιτροπή Ίντα στις 3 Δεκεμβρίου του 2018. Οι διαδικασίες αυτές εξελίσσονται. Τα έγγραφα αυτά είναι προς διαβούλευση και συζήτηση με το Κοινοβούλιο και φυσικά με τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ακολουθούν τη διαδικασία που είχατε προτείνει και εσείς κύριε Λάγκερ το Δεκέμβριο του 16 προς την Επίτροπο Μάλστρομ και την απάντησή της στις 18 Ιανουαρίου του 2017. Ζητούσατε για έναν ρόλο συγκρίσιμο με αυτόν που έχει το Κοινοβούλιο στην επιλογή των δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τα έγγραφα αυτά στην ουσία πραγματώνουν την υπόσχεση της κυρία Μάλστρομ του 17. Λοιπόν, να σας πω ποια είναι τα βασικά σημεία. Καταρχάς, οι υποψήφοι πρέπει να έχουν ε, την ε, υπηκότητα ενός κράτους μέλους, να προτείνονται από τα κράτη-μέλη, ίσως και από την Επιτροπή. Επίσης, μπορεί να είναι και υπήκοοι άλλων χωρών, οι πρόεδροι των ε, δικαστηριών αυτών, των δικαστικών σωμάτων θα προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, αυτές είναι οι προϋποθέσεις σε μια πρώτη φάση για να προταθούν και θα υπάρχει μια μόνιμη επιτροπή επιλογής ανάλογα με τις διαδικασίες για τον διορισμό στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ε, θα πρέπει να είναι υψηλού επίπεδου υποψήφοι, ως δικαστές ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ε, μέλη διεθνών δικαστικών σωμάτων και πάρα πολύ γνωστοί πανεπιστημιακοί. Σύμφωνα με το άρθρο 255 ακολουθείται η διαδικασία για το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ορίζει έναν από τους τέσσερις υποψηφίους που θα αποφασίζονται από την ομάδα επιλογής. Η ομάδα αυτή επιλογής θα ελέγχει τις υποψηφιότητες λοιπόν και θα δημιουργεί μια λίστα υποψηφίων που θεωρείται ότι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι κριτές στα πλαίσια των δικαστικών αυτών ειδικών σωμάτων για τις επενδύσεις. Για κάθε μεμονωμένη συμφωνία θα επιλέγονται πρόσωπα από τον κατάλογο αυτό και αυτό θα συμφωνείτε αλφαγιώτα με την τρίτη χώρα και θα εγκρίνεται από την κοινή ε, επιτροπή η οποία έχει δημιουργηθεί από τη συμφωνία, κάτι που απαιτεί μια απόφαση του Συμβουλίου για να καθοριστεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, χοντρικά αυτή είναι η διαδικασία που περιλαμβάνεται στα έγγραφα τα οποία σας έχουμε στείλει και η διαδικασία μέσω της οποίας θα ορίζονται οι κριτές που θα συμμετέχουν στα ειδικά αυτά σώματα. Έχουμε την αίσθηση ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να διασφαλίσει ότι τα πρόσωπα θα είναι ανεξάρτητα και θα λειτουργούν αντικειμενικά και επίσης θεωρούμε ότι η διαδικασία ε, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, στην ουσία ή μάλλον ε, αντιγράφει τη διαδικασία η οποία έχει ακολουθηθεί τα τελευταία 20-30 χρόνια για το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και θα καταστήσει την επιλογή ανεξάρτητη, αντικειμενική και ισχυρή γενικά και έτσι αναγνωρίζεται και ο ρόλος τον οποίο ζητάτε να αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επιστολή σας του 16. Δεύτερον τώρα για τα ίδια θέματα είναι οι εξελίξεις για το πολυμερές δικαστήριο για τις επενδύσεις. Είχαμε την τρίτη συνάντηση της ομάδας εργασίας η οποία έχει σαν ε, στόχο την μεταρρύθμιση, ε, τις μεταρρυθμίσεις ε, στο δικαστήριο αυτό. Έγιναν συναντήσεις τον Οκτώβριο στην Βιέννη, 19 χώρες ήσαν παρόσες, 400 υποψήφοι, 400 συμμετέχοντες συγγνώμη ήταν επίσης παρόντες, αυτό δείχνει ε, την ε, δυνατότητα σύγκλησης την οποία έχει το σώμα αυτό, ε, την έλλειψη αποκλεισμού ενδιαφερομένων και την αποτελεσματικότητα λειτουργίας μιας τέτοιας οργάνωσης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Και δεύτερον είναι και επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει τη μεταρρύθμιση αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία έχει ζητήσει ε, να γίνονται οι συζητήσει αυτές στο συγκεκριμένο πλαίσιο και αυτά επί τη βάση του ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2015 που ζητά να υπάρξει μια αλλαγή για τα σώματα τα οποία ε, διαμεσολαβούν σε περιπτώσει διαφορών στον τομέα των επενδύσεων, των διεθνών επενδύσεων. Στην ουσία λοιπόν θεωρήθηκε η συνάντηση αυτή τον μήνα Οκτώβριο σαν καθοριστικό σημείο από πολλούς ε, για την μεταρρύθμιση ε, του συστήματος αυτού. Είναι η πρώτη φορά που έχετε ένα πολυμερό σώμα 90 ήσαν οι παρούσες χώρες ε, που κατέληξαν ότι η μεταρρύθμιση του καθεστώτος του ενδιαμέσου αυτού δικαστικού σώματος είναι επιθυμητή. Πρώτον, ζητήθηκε να είναι πιο συνεκτικό το σώμα αυτό, να είναι πιο προβλέψιμο. Δεύτερον, η διαιτητική, η ρόλη η διαιτητική και η ρόλη ενδιαμέσου, όπως επίσης και οι καταστατικές δυνατότητες τις οποίες παρουσιάζει το σώμα αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά τα συμπεράσματα έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ σημαντικά. Η επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας είναι η 1η Απριλίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής θα περάσουμε σε μία συζήτηση ακριβώς για τις επιλογές, τις συγκεκριμένες επιλογές για τις μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πραγματώσουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές την προηγούμενη εβδομάδα στις 19 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη υπέβαλαν δύο έγγραφα προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι διαθέσιμα, είναι στην ιστοσελίδα μας και έχουν αποσταλεί στην Ίντα ε, τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν τις διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν στο μέλλον Εμείς στην ουσία δημιουργούμε το πλαίσιο για την λειτουργία, τη σωστή λειτουργία του πολυμερούς αυτού σώματος. Στην ουσία περιλαμβάνονται οι οδηγίες τις οποίες έχει κάνει δεκτές το Συμβούλιο και το πώς ένα τέτοιο δικαστήριο πολυμερές μπορεί να λειτουργήσει και πώς ένα τέτοιο δικαστήριο για τις διεθνείς επενδύσεις καλύπτει τις ανησυχίες οι οποίες έχουν μέχρι τώρα εντοπιστεί. Είναι σαφές ότι είναι η μοναδική πρόταση η οποία είναι υποσυζήτηση, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες 3.000 πολυμερείς συμφωνίες. Ε, για μας ε, οι τρεις αυτές χιλιάδες συμφωνίες παραμένουν σε ισχύ. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς εμείς θα μεταρρυθμίσουμε τις συγκεκριμένες συνθήκες. Όταν κοιτάμε ακριβώς το τι συμβαίνει, βλέπουμε ότι οι περισσότερες χώρες διατηρούν τις συνθήκες αυτές ή ε, διαπραγματεύονται νέου τύπου. Το CTTPP, σαν παράδειγμα, ε, έχει διάφορες προβλέψεις για την επίλυση των διαφορών, όπως επίσης και η συμφωνία RCEPT, που καλύπτει την Νοτιοανατολική Ασία και την Οκεανία. Από πλευράς μας λοιπόν, εμείς στην ουσία κάνουμε αυτό το οποίο μας ζητήσατε ήδη από το 2016. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας επί τη βάση των ισχυουσών συμφωνιών. Εμείς ε, φυσικά θεωρούμε θετικό αυτό το οποίο αποφασίσατε λίγο πριν για την εμπορική συμφωνία με την Σιγκαπούρη. Ε, είναι ένα σημαντικό βήμα είναι κάτι το οποίο δείχνει την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για τη δημιουργία μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Και είναι κάτι επίσης το οποίο θα διευκολύνει τις σχέσεις με τη Σιγκαπούρη, θα της επιτρέψει να συνεργαστεί μαζί μας για τη δημιουργία ενός πολυμερούς δικαστικού σώματος. Ε, επιταχύνουμε ταυτόχρονα και τις προσπάθειές μας και θα τις επιταχύνουμε για να ενισχύσουμε τη στήριξη για τις προτάσεις οι οποίες κατετέθησαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Θα λάβουμε μέρος σε μια συνάντηση στη Δομινικανή Δημοκρατία με πάρα πολλές χώρες της Κεντρικής Αμερικής για να προωθέσουμε την ιδέα αυτή στα μέσα Φεβρουαρίου ε, θα έρθουμε σε επαφή με ασιατικές χώρες, με αφρικανικές χώρες, με τη Σιγκαπούρη, με τον Καναδά και την Ιαπωνία. Και φυσικά θα επανέλθουμε και μετά από τη συνάντησή μας τον Απρίλιο για να σας μεταφέρουμε τα βήματα προόδου τα οποία θα έχουν μέχρι τότε συντελεστεί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Αρίνα έχει το λόγο λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για, ε, για την ενημέρωση αυτή ε, για το, πολυμερές, ε, για το Πολυεθνικό Δικαστήριο, μάλλον το ΜΙΚ, είχε υποβληθεί μια ερώτηση στο 10 για το ICS στο πλαίσιο ΣΕΤΑ από το Βασίλειο του Βελγίου. Κανονικά πρέπει να έχουμε μια ερώτηση από το δικαστήριο φέτος. Πώς θα ενσωματώσετε λοιπόν την απάντηση του δικαστηρίου στη συμφωνία της Σιγκαπούρης για παράδειγμα που ψηφίστηκε σήμερα ως προς τις προσαρμογές που ενδεχομένως θα χρειαστούν σε σχέση με την απάντηση του δικαστηρίου. Βρίσκω, πιστεύω, ότι να έχουμε μια διάταξη ήδη εγκατεστημένη αλλά που θα μπορούσε να έχει κάποιες περιπλοκές ή δυσκολίες λόγω της απάντησης του δικαστηρίου πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, πώς σκοπεύει η Κομισιόν να διαχειριστεί το ζήτημα όταν θα έχουμε την απάντηση του δικαστηρίου. Σας ευχαριστώ κυρία αλλά έχει λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομισιόν για την έκθεση αυτή. αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξε ιδιαίτερη προσοχή από κάποιες χώρες για το ζήτημα αυτό. Αναφέρθηκε η Ινδία και η Νότια Αφρική. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να ξέρουμε ποια θα ήταν η συνεισφορά των χωρών αυτών και αν θα, υπήρξε, θα υπήρχε αντίκτυπος για το αποτέλεσμα. Η Νότια Αφρική υπήρξε ένας από τους ηγέτες ε, για τις δεσμευτικές αυτές διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γενέβη. Ίσως λοιπόν να ανησυχούσε μια τέτοια χώρα για την ε, επικυρίαρχη θέση των επενδυτών έναντι των πολιτών. Επίσης το όριο της συμμετοχής προκειμένου να προχωρήσουμε επιτυχώς ε, προς την σύμβαση ΜΙΚ. Τι ακριβώς εννοείται με αυτήν την διατύπωση. Η κυρία Μινό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι, Πρόεδρε, που η Κομισιόν βρήκε το χρόνο να έρθει να μας πει για τις εξελίξεις σχετικά με το δικαστήριο, το πολυμερέγγις δικαστήριο το επενδυτικό. Την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν μάλιστα υπέβαλε και μια πρόταση σχετικά με τον μηχανισμό αυτών επίλυσης ε, κρατικών διαφορών. χιλιάδες πολίτες υπέγραψαν μία μία αναφορά που προσπαθούν να σταματήσουν το ICS. Επομένως οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά το ζήτημα. Στη Βιέννη ετέθε ένα ερώτημα σχετικά με τους ε, υπευθύνου του δικαστηρίου, δηλαδή αυτούς που θα είναι υπεύθυνοι για την επιμήλυση των διαφορών. Όλα αυτά όμως ε, ε, τα σπρώξαμε υπό τα διάφορα και δεν ε, τύχανε μεγάλης προσοχής. Η Κομισιόν με όλα αυτά τι σκοπεύει να κάνει, γιατί είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και για εμάς και για τους πολίτες. Υπάρχει και ένα ακαδημαϊκό φόρουμ το οποίο υποτίθεται ότι θα συγκατευθύνει υποτίθεται το ICS κάποια μέλη του οποίου είναι και μέλη των αντιπροσωπείων το οποίο δεν φαίνεται καθόλου κατάλληλο. Ως προς αυτό τι έχει να πει η Κομισιόν. Επίσης, οι εθνικές δικαστικές οδοί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί το να τοποθετούμε όλα αυτά τα ζητήματα υπό τα διάφορα μου φαίνεται πραγματικά παράδοξο. Γιατί αν δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο ούτε το εθνικό δίκαιο μου φαίνεται υπερβολικό. Και ποια θα είναι η σχέση μεταξύ του πάνελ και του ευρωπαϊκού δικαίου. Οπωσδήποτε το, το ΔΕΚ θα πρέπει να έχει το τελευταίο λόγο εδώ. Ο Παύλος Ρίμπιχ έχει το λόγο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ε, πώς βλέπετε τη διαφορά ή τη σχέση ανάμεσα στους ε, κανόνες ε, του WTO του και ε, το δευτεροβάθμιο όργανο, καθώς με τις ε, ε νέες εξελίξεις ε, ουσιαστικά δεν είναι δυνατή η επίλυση των διαφορών σε τεχνικό επίπεδο αλλά όλα περνάνε στο στρατιωτικό επίπεδο και το ίδιο συμβαίνει βέβαια και σε διμερές επίπεδο, σε διμερές συμφωνίες δηλαδή όταν δεν υπάρχει κανένας ο οποίος μπορεί να είναι αρμόδιος για τη λήψη μιας απόφασης ε, τότε και πάλι ε, επιβάλλεται η βία. Και η επιβολή βέβαια τη ε, βία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απορρίπτουμε σε μια δημοκρατία. Θα πρέπει να είμαστε υπέρ τη ελληνική επίλυση διαφωνών και γι' αυτό νομίζω πω η Επιτροπή θα πρέπει να επιμείνει στην ύπαρξη τέτοιων μηχανισμών. Γιατί είδαμε, για παράδειγμα, τι συμβαίνει σε περίπτωση εμπορικού πολέμου με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τους ε, κινητήρες και το καθεξής, ε, ουσιαστικά εκείνοι που υπέστησαν ε, τις συνέπειες ήταν εργαζόμενοι και είναι πραγματικά εκεί ήταν πολύ ορατή η έλλειψη ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Θα πρέπει λοιπόν οι διεθνείς οργανώσεις και οι διεθνείς θεσμικά όργανα πάντοτε να βρίσκουν τέτοιου είδους λύσεις που να οδηγούν δηλαδή στην ελληνική επίλυση των διαφορών. Από δικής μου πλευράς προερχόμενο από το βορρά της Γερμανίας, προφανώς έχω τεράστια υπομονή, λέει ο πρόεδρος. Αλλά εν ώψη όλων αυτών στοιχείων ε, την έχασα. Αυτά τα τρία βήματα τα συζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για όλες τις ανησυχίες και οι ανησυχίες για το ISDS έχουν εκφραστεί πάρα πολύ καιρό τώρα. Ε, εγώ δεν κατανοώ γιατί χρειάζεται τόσο πολύς χρόνος. Το είχαμε συζητήσει και στα πλαίσια της TTIP. Ήταν σαφές. Άρα τελικώς η ερώτηση είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι αποδεκτό. Είναι αποδεκτό να μας χρειάζονται τρία χρόνια για να μεταρρυθμίσουμε κάποια απλά στοιχεία. Και ποιος είναι τελικός υπεύθυνος. Υπάρχουν κράτη-μέλη, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που προσπαθούν να υποσκάψουν αυτήν την απαραίτητη διαδικασία και πλαισίωση. Και αν δεν έχουμε αποτέλεσμα στο άμεσο μέλλον, δεν θα ήταν καλύτερο απλώς να εστιαστούμε στο ευρωπαϊκό μας πλαίσιο και τίποτε άλλο. Um, um, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, τα σχόλια. Αν μου επιτρέπετε θα τα διατρέξω κατά σειράν, λέει ο μιλητής, για την ερώτηση της κυρία Αρενά. Ναι, υπάρχει η ερώτηση προς το ΔΕΚ σχετικά με τη συμβατότητα του επενδυτικού δικαστηρίου με την ευρωακή νομοθεσία. Περιμένουμε την ε, γνωμοδότηση στις 29 του μηνός, μάλλον της ε, εισαγγελίας και του δικαστηρίου σύντομα μετά. Πάντω έχουμε σχεδιάσει προσεκτικά το SDS ώστε να είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχε πει ότι και το σύστημα ΣΕΤΑ ήταν συμβατό. Πρέπει να περιμένουμε τώρα να δούμε τι τελικός, πώς τελικός θα τοποθετηθεί το ΔΕΚ. Εάν το ΔΕΚ θεωρήσει παρόλες αυτές τις προσπάθειες ότι υπάρχει ασυμβατότητα, τότε κατά τις εβραϊκές συνθήκες ή οι σχετικές συνθήκες της Σιγκαπούρης και η ΣΕΤΑ δεν θα μπορέσουν να τεθούν ισχύ μέχρι ότου θα έχει επιληθεί το ζήτημα αυτό. Ε, όπως γνωρίζετε η ΣΕΤΑ αυτή τη στιγμή επικυρώνεται από τα Εθνικά Κοινοβούλια και για την IPA της Σιγκαπούρης εφόσον την εγκρίνει η Ολομέλεια, θα πρέπει επίση να επικυρωθεί από την Εθνικά Κοινοβούλια. Θα χρειαστεί λοιπόν χρόνος μέχρι, να τεθούν σε ισχύ οι συμφωνίες αυτέ. Εάν το ΔΕΚ τοποθετηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, τότε θα πρέπει εμείς να κινηθούμε προκειμένου να διορθώσουμε πριν τη θέση σε ισχύ. Δεν θα μπορούσα τώρα να πιθανολογήσω για το τι θα πει το ΔΕΚ. για τις ερωτήσεις της κυρίας Χάουταλα. η όλη η προσέγγιση είναι συμμετοχική. Έχουμε 90 χώρες που ενέχονται, η Νότιος Αφρική είναι μία από αυτές, ε, συνομιλούμε συχνά με τους νότιοαφρικανούς ε, συναδέλφους, ομολόγους, έχουν ε, επιδείξει ενδιαφέρον για την μεταρρύθμιση συνολικά έχουν δείξει ενδιαφέρον για τις ιδέες που έχουμε υποβάλει και έχουν μια περίοδο χρονική εντός της οποίας μπορούν και εκείνοι να υποβάλουν προτάσεις και συνεισφορά στη συζήτηση. Δεν έχω κάποιες ενδείξεις σήμερα ότι θα το πράξουν αυτό, αλλά εάν το πράξουν, οπωσδήποτε θα είναι και αυτό μέρος της όλης ε, συζήτησης του όλου διαλόγου και για τα όρια Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε μία ψήφο ενώπιον της Ολομελίας των Ηνωμένων Εθνών και το έργο της Σατράλ θα έπρεπε να το εγκρίνει ακριβώς η Ολομέλεια και εφόσον το εγκρίνει θα πάμε στην σύσταση του Πολυμερούς Επαθητικού Δικαστηρίου Και εκεί πρέπει να δει κανεί πόσε χώρε πρέπει να προσχωρήσουν προκειμένου ο μηχανισμό να είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή είναι να λειτουργεί ομαλά. Δεν είμαι βέβαιο για αριθμό αυτό, αλλά πρέπει να είναι στην τάξη μεγέθου 40 ή 50. Τώρα η διαδικασία του Σατράλ και έχει επιμείνει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή στο να λάβει υπόψη τη όλες τις ανησυχίες που εκφράζονται εστιάζεται ακριβώς σε ανησυχίε επί της διαδικασία. και μπορούμε να δούμε και άλλα δυνητικά θέματα και η χρονική στιγμή είναι τώρα για να δούμε πώς αυτά θα μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. Αναφερθήκατε στο ρυθμιστικό ζήτημα που και εμάς μας ανησυχεί αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι μέσω της δημιουργίας ενός τακτικού σώματος, μόνιμου σώματος, γιατί αυτές οι ατάξεις τις, τις βρίσκουμε και στα εθνικά συστήματα τα νομοθετικά. Δεν είναι οι διατάξεις που είναι το πρόβλημα, αλλά είναι οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ένα μόνιμο σώμα. Αναφερθήκατε επίσης στο Ακαδημαϊκό Φόρουμ και στους διαμεσολαβητές. Είναι απολύτως σαφές ότι στην διαδικασία Ονσατράλ ότι η εντολή της είναι κρατική Ε, ε, το λέγει ξεκάθαρη παράγραφος 10 της διαδικασίας και το καθιστούμε 100% σαφές ότι οι αποφάσεις πολιτικής στην Ουστατράλ λαμβάνονται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων που έχουν την κατάλληλη εντολή από τις πολιτικές τους ηγεσίε, στην περίπτωσή μας και το Συμβούλιο και αυτήν εδώ την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά. Μιλούμε λοιπόν για αξιωματούχους των κυβερνήσεων που λογοδοτούν στα κοινοβούλια και στις νομοθεσίες τους. Η παρουσία των διαμεσολαβητών είναι κάτι που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο κοιτώντας, εξετάζοντας τεχνικά ζητήματα. Οι αποφάσεις όμως οι πολιτικές θα λαμβάνονται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων. Και στην ερώτησή σας γιατί δεν υπαρκεί η εθνική νομοθεσία είναι αντίστοιχο με αυτό που είπε ο κύριος Ρούμπιχ. δουλεύουμε εδώ και καιρό σε επενδυτική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στο γεγονός ότι η κινέζικη δικαιοσύνη θα σεβόταν τις ε, δικές μας νομοθετικές διατάξεις και δυστυχώς το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τις ε, αμερικανικές αρχές. Εξού και δεν θεωρούμε επαρκή την ε, εθνική νομοθεσία και το εθνικό πλαίσιο δικαιοσύνης. Μιλούμε για διεθνείς συμβάσεις και δεσμεύσεις. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσει κανείς ότι ο μηχανισμός αυτός που έχουμε υποβάλει, που έχουμε επιτάπητο, έχει μια ανοιχτή ρήτρα δικαιοδοσίας. Τεχνικώς αυτό σημαίνει ότι όπως εξελίσσονται συν το χρόνο οι συνθήκες, εφόσον ληφθούν οι αποφάσεις, και αυτό έχει ήδη συμβεί σε κάποιες, να προσθεθούν υποχρεώσεις για τους επενδυτές, το πολυμερές δικαστήριο μπορεί να αναλάβει την εξέταση αυτών των θεμάτων. Και για τις ερωτήσεις του κυρίου Ρούμπιχ, αντιλαμβανόμαστε απολύτως ε, και είναι η ίδια ομάδα που ασχολείται με το σώμα προσφυγών του ΠΟΕ, κάποια από τα διδάγματα εμφανίζονται στο έγγραφο στο οποίο αναφέρθηκα. Δηλαδή, καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να μπλοκάρει το διορισμό των δικαστικών. Και δεν θα υπάρχει αυτό το θέμα της ανανέωσης της θητείας τους, που είναι στη βάση της κρίσης στο σώμα προσφυγών του ΠΟΕ. Και όπως γνωρίζετε, ε, χρησιμοποιούμε στις διμερείς συμφωνίες μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Η Συμφωνία της Κορέας είναι ένα παράδειγμα της Ουκρανίας για τις ε, περιορισμούς εξαγωγών ξυλίας είναι άλλο ένα παράδειγμα. Και τέλος κύριε Λάγκα, πράγματι έχει χρειαστεί χρόνος, συμφωνώ μαζί σας, έχει πάρει χρόνο η προσπάθεια αυτή. Από την άλλη μεριά, όπως είπα από την αρχή, είναι η πρώτη ενδελεχή συζήτηση που λαμβάνει χώρα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, πολυμερές επίπεδο και αυτό που συνειδητοποιούμε είναι ότι ενώ καθότι οι ανησυχίε, μάλλον την ώρα που οι ανησυχίε αυτές που υποβάλλονται, εκφράζονται, είναι προφανείς για εμάς και εκφράστηκαν το 2014 και το 2015 για την TTIP, πολλές άλλες χώρες δεν έχουν φτάσει, αν θέλετε, στο προκεχωρημένο στάδιο ανάλυσης που έχουμε φτάσει εμείς και νομίζω ότι η διαδικασία αυτή είναι ακριβώς πάρα πολύ χρήσιμη προκειμένου να προσελκύσει και άλλους συνομιλητές και να δεχθούν το συμπέρασμα ότι η συστημική μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη. Εν είχαμε θέσει τα ερωτήματα αυτό το 2014-2015 κανείς δεν θα είχε προσέλθει στο τραπέζι της συζήτησης. Και πράγματι χρειάζεται χρόνο, αλλά με τη σταδιακή αυτή προσθήκη συνομιλητών εταίρων αναφερόμαστε σε αυτό το πλαίσιο των 3.000 συμβάσεων στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα. Θα δούμε ποιες επιλογές θα τεθούν ακόμα και τελικώς η ομάδα εργασίας θα πρέπει να φασίσει ποιες από αυτές τις επιλογές θα είναι εκείνες στις οποίες μπορεί να βασιστεί. και αν αυτές συμπεριλαμβάνουν το πολυμερές δικαστήριο το επενδυτικό, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Συζητούμε με τους εταίρους και με την γραμματεία Central μηχανισμούς για να επιταχύνουμε τη δουλειά, να έχουμε ενδιάμεσες συναντήσεις, παρατάσεις συναντήσεων κτλ. Ε, το χρονικό ζήτημα πάντως το έχουμε λάβει υπόψη. Ε, ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας και διμερώς να απαντήσουμε ακόμα περισσότερες. Εκόλυν, λέει ο πρόεδρος. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ζητούν όλοι οι εταίροι στα Ηνωμένα Έθνη τέτοιο είδους μηχανισμό. Ω προ το ISDS ήταν κυρίω οι χώρε οι ευρωπαϊκέ και οι Ηνωμένε Πολιτείε που το ζητούσαν. Εφόσον εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια σαφής αντίληψη των ανησυχιών των πολιτών και μια πρόθεση μεταρρύθμισης, τότε οι χώρες που ζητούν ένα τέτοιο μηχανισμό θα έπρεπε να είναι να ηγούνται τις προσπάσεις μεταρρύθμισης. Ανεξαρτήτως των απόψεων των υπολείπων χωρών. Και δείτε την περίπτωση της Σιγκαπούρης. Η Σιγκαπούρη δεν ζήτησε το επενδυτικό κομμάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτησε. Και ευτυχώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να πείσει Κομισιόν και Συμβούλιο ότι χρειαζόμαστε ένα δημοκρατικό σύστημα. Έναν ανεξάρτητο δηλαδή φορέα δικαιοσύνη. Αρχικά η Κομισιόν ζητούσε από τη Σιγκαπούρη το κλασικό ESDS. Επομένω υπάρχει πολύ συγκεκριμένη ευθύνη για τι χώρε εκείνε που έχουν το συμφέρον και το ενδιαφέρον να ζητούν τέτοιους μηχανισμούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτηματά και να κάνω κάποιες παρατηρήσεις μετά από τα όσα ακούσαμε, κύριο εκπλήσωμε πραγματικά γιατί αν θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε να περιορίσουμε το ρεγκλατόρ, τότε τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να μην έχουν τόσο μεγάλη πρόσβαση οι εξωτερικοί επενδυτές δηλαδή. αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με το ISDS, ότι δηλαδή δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θα έπρεπε. Και ε, ε, εδώ δεν αναφέρομαι μόνο στο διεθνές δίκαιο, αναφέρομαι και στο ενωσιακό δίκαιο, αλλά και στο ε, εθνικό δίκαιο, στο περιφερειακό δίκαιο. Όλα αυτά λοιπόν, σε όλα αυτά τα επίπεδα υπάρχει δυνατότητα πλέον προσβολής αυτών των νομοθεσιών. Οπότε, αν ε, έχουμε όλες αυτές τις ε, η, δική σας προσέγγιση είναι, ε, είναι αυτή, αλλά διαρωτώ με κατά πόσο είναι σωστή. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο ε, είναι σωστή αυτή η βάση όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις άμερες ξένες επενδύσεις και την, ε, τους σχετικούς μισθούς οι οποίοι θα θα διασφαλιστούν αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πρόκειται για έναν τρόπο με τον οποίο προωθούμε την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούμε θέσει εργασία. Δηλαδή, ε, είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε όλοι. Πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι. Δεν μπορούμε δηλαδή να αντιμετωπίζουμε ευνοϊκότερα του ε, ε, είμαι μεταπούς αν θέλετε επενδυτές σε σύγκριση με τους αλλοδαπούς ε, επενδυτές οπότε ε, πραγματικά θεωρούμε πως είναι καλή αυτή η προσέγγιση της Επιτροπής για να βρούμε μια λύση δηλαδή χωρίς να είναι ανάγκη, ε, αναγκαία μια στρατιωτική παρέμβαση. Ο Κόλλιν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ για αυτά τα συμπληρωματικά σχόλια. σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, να σας πω πως η διαδικασία είναι πραγματικά εντυπωσιακά ανοιχτή. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο αριθμό ε, εγκεκριμένων παρατηρητών, μη κυβερνητικέ οργανώσει, συνδικαλιστικέ οργανώσει, οργανώσει των πολιτών. Οπότε μπορούν όλοι αυτοί οι παρατηρητέ να παρακολουθήσουν τι συζητήσει, να συμμετάσχουν στι συζητήσει. Υπάρχουν ε, και μαγνητοφωνημένε αυτέ οι συζητήσει ε, και πλήρε εκθέσει οι οποίε καταρτίζονται μέσα σε χρονικό διάστημα μία εβδομάδα από την κάθε συζήτηση. Οπότε ίσως κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλά αντίστοιχα παραδείγματα διαφάνειας ε, όπως ε, το συγκεκριμένο και πραγματικά είναι κάτι το οποίο εκτιμά η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αυτό το επίπεδο διαφάνειας. Ε, τώρα, απαντώντας στο ερώτημά σας κύριε Λάγκη. Ναι, προφανώ θα πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία. και θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν διμερείς συμφωνίες επενδύσεων ε, ε, σε αριθμό 1.400 που έχουν εγκριθεί από τα διάφορα κοινοβούλια τα τελευταία 30 με 40 χρόνια. Πολλές από αυτές τις συμφωνίες είναι παλιές, είναι παροχημένες και τις οποίες θέλουμε να αναθεωρήσουμε. Θέλει και το κοινοβούλιο να τις αναθεωρήσει και τα κράτη-μέλη θέλουν να τις αναθεωρήσουν ώστε να ανταποκρίνονται στα πρότυμα που έθεσε το κοινοβούλιο στο ψήφισμά του του 2015. Εάν λοιπόν θέλουμε να το επιτύχουμε αυτό και έχουμε τόσο υψηλό αριθμό συμφωνιών, τότε χρειαζόμαστε μια διαδικασία η οποία όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή και στην οποία συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερε χώρε, ώστε να καταλήξουμε στο κατάλληλο εργαλείο, στο κατάλληλο μηχανισμό. Ε, και εγώ βέβαια εκνευρίζομαι το γεγονό, όπω και εσεί, ότι η διαδικασία δεν τρέχει ταχύτερα, αλλά αυτή είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Εμεί από την πλευρά τη Ένωση ασκούμε πιέσει και έχουμε βασιστεί συστηματικά στη Σιγκαπούρη, στον Καναδά και σε άλλες ε, χώρε οι οποίες ασκούν και εκείνες πιέσεις. Πάντω εκείνο που δημιουργεί έκπληξη σε σχέση με αυτές τις ε, ε, συνομιλίε. είναι το γεγονός ότι πολλέ άλλες χώρες με τις οποίες δεν έχουμε άμεσες σχέσεις, δηλαδή δεν έχουμε μια άμεση συμφωνία IPA ή συμφωνία FTA και εκείνε τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ μια αναθεώρηση. επανερχόμενο τώρα στο ζήτημα που έθεσε η κυρία ε, Μινέο σε ό,τι αφορά την ουσία του θέματος. Η πραγματικότητα είναι, όπως σα είπα, ότι έχουμε 3.000 τέτοιε φωνές οι οποίε. Ε, ανα, τυχάνουν συνεχούς αναδιαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα, η Κορέα αυτή την περίοδο ε, διαπραγματεύεται μια νέα συμφωνία ε, που περιλαμβάνει ISDS. Υπάρχει μια νέα ε, διαβούλευση ό,τι αφορά το ICPPT. Ε, νέα διαβούλευση έχει ξεκινήσει και μεταξύ των ασιατικών χωρών. Σε όλε αυτέ τις συμφωνίε και πάλι περιλαμβάνεται πάντοτε το ISDS. Και εδώ, περνάω σε αυτό που ανέφερε ο κύριο Ρούβικ, θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να αφήσουμε δηλαδή τους ξένους μας επενδυτές χωρίς καμία προστασία ενώ οι ανταγωνιστές μας από την Αμερική, από την Κίνα και οπουδήποτε αλλού τους παρέχουν προστασία ή θέλουμε αντιθέτως να τους παράσουμε την κατάλληλη προστασία διασφαλίσοντας όμως ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει υπερβολική, υπερβολικό, υπερβολικός κανονιστικός αν θέλετε ε, ε, φόρτος. Ε, εκείνο νομίζω που λοιπόν που θα πρέπει να κάνουμε είναι ε, να ε, προβλέψουμε αυτές τις αναθεωρήσεις με τον κατάλληλο τρόπο τους ώστε να μην προβλέψουμε υπερβολικά πολλούς κανόνες που θα διέπουν αυτές τις εμείς. Ευχαριστώ. Λέω ο Πρόεδρο, το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι μια, ένα περίπλοκο ζήτημα αυτό και δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε, να το εξετάσουμε στο σύνολό του. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο τη σημερινής διάταξη, το σημείο 30, δηλαδή τι διαπραγματεύσει στο πλαίσιο μια συμφωνία Ελεύθερο εμπορίο με την Ινδονησία που ξεκίνησαν οι εν λόγω συνομιλίες για την εν λόγω συμφωνία τον Ιούλιο του 2016. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι το εξαιρετικά ε, πρόσφατο. Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια κυρία Χέλενα Κιούνικ βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας που είναι η κύρια αρμόδια για τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο αυτής ε, της ε, μελλοντικής συμφωνίας με την Ινδονησία. Οπότε τη δίνω το λόγο για πέντε λεπτά για να μα ενημερώσει ω προς το πού βρισκόμαστε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. σα ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει με την Ινδονησία ε, και επιτρέψτε μου καταρχήν να σα θέσω ένα γενικότερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μα με την Ινδονησία. Θα θυμόσαστε ότι η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη χώρα της Ασίας ε, και ε, εκπροσωπεί το 36% των χωρών της ΑΣΕΑΝ ε, με πληθυσμό 250 εκατομμυρίων. Και σημειώνει κατά τελευταία χρόνια μια εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα η Παγκόσμια Τράπεζα προέβλεψε ότι έως το 2030 ενδέχεται η Ινδονησία να είναι η 7η ε, ισχυρότερη, αν θέλετε, οικονομική δύναμη, η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Άρα λοιπόν υπάρχουν όλε αυτέ τι θετικέ προοπτικέ, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και μία σειρά από πολύ σημαντικέ προκλήσει προκειμένου να ξεφύγει από τη φτώχεια η εν λόγω χώρα. Ακριβώς ε, και επειδή υπάρχει αυτός ο πολύ μεγάλος ε, αριθμός ε, κατοίκων, η αύξηση της μεσαίας τάξης, η αύξηση Τη ε, αστιφιλία που δημιουργεί και αυτή ε, τι δικές της πιέσει ε, και επίσης υπάρχει μεγάλη ανάγκη επενδύσεων στον τομέα της, του λιανικού εμπορίου, των νέων τεχνολογιών και εδώ βλέπουμε και πολλές ευρωπαϊκές εταιρείε οι οποίες δραστηριοποιούνται σε μια σειρά από κλάδους. Και πλέον να, να, επίσης να πω ότι οι οικονομίες μας είναι συμπληρωματικές και υπάρχει ένα δυναμικό αναξιοποίητο ακόμα σε μια σειρά από ε, δηλαδή είναι ο πέμπτος κατά σειρά εμπορικό μα εταίρο ε, μεταξύ των χωρών τη ΑΖΕΑΝ και αυτό καταδεικνύει από μόνο του πόσε δυνατότητε ακόμα υπάρχουν. Ε, έχουμε συμπεριλάβει κάποιε όχι τόσο ευαίσθητε, αν θέλετε, ευαίσθητου τομεί όπως είχαμε σε σχέση με άλλους όπως την Αυστραλία, δηλαδή σε ό,τι αφορά το βόλιο κρέα και άλλα αγροτικά προϊόντα, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν κάποια ε, ακόμα αγαθά ε, στα οποία θα επανέλθω. Και ακόμα να πω ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ε, βήμα, αν θέλετε, αυτή η συμφωνία με την Ινδονησία σε ό,τι αφορά την εδραίωση τη θέση μα στι χώρε τη ΑΣΕΑΝ, τόσο μέσο όσο και μακροπρόθεσμα. Και επίση πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προκειμένου να θεμελιώσουμε και να εδραιώσουμε, αν θέλετε, την εντάξει με βάση του κανόνε οι οποίοι έχει τεθεί ένα αμφιβόλο τελευταία χρόνια. Τώρα, έρχομαι στι ίδιε τι διαπραγματεύσει. εξελίσσονται, αλλά ε, με αργούς ρυθμούς και αυτό ε, οφείλεται σε μια σειρά από, από λόγους. Καταρχήν υπάρχουν ε, πολλοί περιορισμοί στην οικονομία της Ινδονησίας που προέρχονται από την ιστορικά εξαιρετικά προστατευτική στάση που τηρεί η χώρα αυτή. Και εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε και το οποίο συμφωνήθηκε κατά το scoping exercise είναι να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια όσο το δυνατόν πιο ευρεία συμφωνία με την Ινδονησία, την ευρύτερη που θα έχει υπογράψει μέχρι στιγμή. Οπότε υπάρχουν μια σειρά από προκλήσει, θα χρειαστούν μια σειρά από αλλαγέ στην νομοθεσία, ε, προκειμένου να συναυθεί η συμφωνία. Και επίση, ε, ένα ακόμα ζήτημα που περιπλέκει τα πράγματα είναι το γεγονό ότι επίκυνται το, μέσα τώρα, στον Απρίλιο δηλαδή του 2019, προεδρικέ εκλογέ. Οπότε σε μια χώρα τόσο τεράστια όσο η Ινδονησία υπάρχουν μια σειρά από θέματα που περιπλέκουν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά έχουμε επιτύχει κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μας ε, πρόσφατα. Συμφωνήσαμε ε, καταλήξαμε συμφωνία ε, ε, με, την ΕΦΤΑ και με την Αυστραλία. αλλά ακόμα δεν έχει γίνει υπογραφή λόγω κάποιων εκκρεμωτήτων ακόμα που έχουν προκύψει. Αλλά και πάλι δεν έχουμε κινηθεί μέχρι εκεί που θα θέλαμε. Τώρα, υπάρχει ένα είναι το φινικέλαιο, ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα, παρότι όπως σας είπα τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα δεν είναι τόσο προβληματικά. Ε, και, ε, έχουμε ξεκινήσει και μια διαδικασία ξέρετε, συγκεκριμένα του φινικελαίου και της βιώσιμης, βιωσιμότητας δηλαδή της παραγωγής του Ε, ναι, και θα πρέπει ε, στο πλαίσιο της ε, διαδικασίας απορρίθμισης την οποία ακολουθούμε να δούμε πώς θα εντάξουμε και αυτές τις αγωγές. Σε ό,τι αφορά το φινικέλαιο, να πούμε ότι η Ινδονησία συμφωνεί ως προς το ότι ναι, το, το, η βιωσιμότητα του φινικελαίου θα πρέπει να είναι διασφαλισμένη. Απλώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι τα κριτήρια τα οποία θα ορίζουν αυτήν τη βιωσιμότητα. Γιατί δεν υπάρχει μια διεθνή συμφωνία ως προς αυτά τα κριτήρια, ούτε υπάρχουν και σχετικοί κανονισμοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω για παράδειγμα συμβαίνει στο επίπεδο τη ξυλία. Άρα λοιπόν μιλάμε για διαπραγματεύσει οι οποίε συνεχίζονται, συνομιλίε οι οποίε θα ξακολουθήσουν για κάποιο χρόνο ακόμα. Πάντω, προτού προβούμε στη σύναψη οποιαδήποτε συμφωνία, θα πρέπει να φτάσουμε σε κάποιο είδο λύση έτσι ώστε η σχετική παραγωγή να είναι βιώσιμη. Και κάτι τέτοιο βέβαια θα είναι προ το συμφέρον και τη ίδια τη συντονισία και θα δούμε πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα όταν θα περάσουμε σε αυτό. Ε, δεν λέμε ότι ε, δεν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, αλλά προς την πλευρά είναι ένα είδος ε, κινητού στόχου, δηλαδή παραμένει δύσκολο. Τώρα, ο επόμενο γύρο διαπραγμάτευσης θα λάβει χώρα εδώ, στι Βρυξέλλες, και στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν συζητήσει σε σχέση με όλα τα επιμέρου κεφάλαια τη συμφωνία. Θα εμβαθύνουμε τη συζήτησή μα σε ό,τι αφορά ε, την, ε, την προσφορά που κάναμε ε, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις, όπως δηλαδή αυτή είχε υποβληθεί κατά τον έκτο γύρο διαπραγμάτευσης και επίσης θέλουμε να επιτύχουμε κάποια περαιτέρω πρόοδο σε ό,τι αφορά τι κρατικέ συμβάσει. Μέχρι στιγμή δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση η Ινδονησιακή πλευρά. Αλλά θα δούμε από εδώ και μετά ε, πότε ακριβώς θα ανταλλάξουμε τις ε, ε, προσφορές μας και πώς θα κινηθούμε από εκεί και μετά ούτως ώστε να ξεκινήσουν και οι διαπραγματεύσεις εδώ. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ε, όλοι οι λόγοι για τους οποίους ξεκινήσαμε αυτές τις διαπραγματεύσεις το 2016 εξακολουθούν να ισχύουν. Πρόκειται για περίπλοκε διαπραγματεύσει, οι οποίε δεν κινούνται γρήγορα, αλλά στι οποίε επιτυχάνουμε σταθερή πρόοδο σε σχέση με όλα τα κεφάλαια τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και βλέπουμε να υπάρχει ενδιαφέρον από την Ινδονησιακή πλευρά. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση παραμένει περίπλοκη για εκείνους, όπως είπαμε, τόσο λόγω του συστήματος το οποίο ισχύει ιστορικά εκεί, αλλά λόγω και των επικείμενων προεδρικών εκλογών. Εάν καταφέρουμε να καταλήξουμε στη σύναψη μιας συμφωνίας, σίγουρα θα ήταν κάτι το ε, θετικό, όχι σε ό,τι αφορά μόνο την πρόσβαση στην αγορά, αλλά και σε ό,τι αφορά την εδραίωση ενός συστήματος ε, κανόνων, ε, σε σχέση με μία από τις σημαντικότερες χώρες της ΑΣΕΑΝ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή μας, τον κύριο Μάρτιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Κόνιν για την παρουσίασή της. Μετά τη Σιγκαπούρη λοιπόν και ελπίζουμε και το Βιετνάμ τους επόμενους έξι μήνες, η Ινδονησία θα είναι το επόμενο κομμάτι στο πάζλ των ασιατικών χωρών δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε βέβαια. Υπάρχουν πολλά και ευαίσθητα θέματα και το βασικό είναι το φινικέλαιο. Ένας μεγάλος αριθμός μικιό ανησυχούν γιατί οι διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία δεν θα αλλάξουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά μπορούν να να αποδυναμώσουν τις διακανονιστικές οδηγίες και ρυθμίσεις και γι' αυτό ε, κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβεί φυσικά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε επίσης ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι συμβατές με τις ε, ε, αποφάσεις του ΠΟΕ και δεν θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ινδονησία να προσφύγει στον ΠΟΕ. Indonesia has ratified all the core ILO conventions. Σχετικά με το ESD, ε, κάποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί από πλευράς της Ινδονησίας, είναι θετικό, αλλά η εφαρμογή έχει μείνει πίσω. και τελικά θα πρέπει να έχουμε και ένα μηχανισμό σε σχέση με τα TSD κυρώσεων όπως και με τους Σιγκαπουριανούς θα πρέπει και οι Ινδονήσοι να έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν σε ένα τέτοιο μηχανισμό για το TSD. Ε, τώρα σχετικά με τα ενδιάμεσα δικαστικά σώματα ε, ε προφανώς ε, είναι προφανής η απόφαση των Ινδονησίων να διακόψουν την ε, την λειτουργία μάλλον όλων των ε, ε, ενδιάμεσων διατητικών σωμάτων. Αλλά επαναλαμβάνω προβλήματα όπως το φινικέλαιο, η αποψήλωση των δασών και άλλα γεωργικά προϊόντα οδηγούν στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και της πανίδας επίσης υπάρχουν πάρα πολλά ε, πρωτεύοντα θηλαστικά τα οποία θα απειληθούν. Ταυτόχρονα αυξάνεται η θέση της ε, Ινδονησίας ως από τις βασικές χώρες εξαγωγές ε, βατράχων προσβρώση. Ξέρουμε ότι κυριαρχεί στην αγορά αυτή η Γαλλία. Ε, είναι λοιπόν λίγο περίεργο λόγω αυτής της ενδενησίας, ε, της ευαισθησίας συγγνώμη, της συνδονησίας δεν προτείνουμε κάποια μέτρα αντίστοιχα με αυτά τα οποία είχαμε προτείνει στο Μεξικό και στο Βιετνάμ και διαρωτώ αν μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στις διαπραγματεύσεις μας σε σχέση με το θέμα της προστασίας της πανίδας Θα δώσω τώρα το λόγο στους Κιώδης. Ο κύριος Ζαντό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποια μέρα θα συζητήσουμε το θέμα της γαστρονομίας. Και κινδυνεύει να είναι αρκετά σενιό το θέμα αυτό με αίμα δηλαδή λίγο ψημένο τώρα ε, το βασικό, ένα από τα βασικότερα θέματα της συζήτηση αυτής είναι πράγμα το φινικέλαιο μέσω της ΦΛΕΚΤ ε, το κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια ε, είχε επιχειρήσει καθότι η Ινδονησία ε, παραμένει μια χώρα στην οποία η υλοτομία και η δασοκομεία γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών να θέσει να μπορέσει να προσεγγίσει το θέμα αυτό. Όταν στο παρελθόν ο πρόεδρος Μπαρόσο είχε πάει στον Καναδά για να γιορτάσει μαζί με τον Στίβεν Χάρπερ ε, την ΣΕΤΑ, ε, την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αλλάξει γραμμή ε, για τις κυρώσεις που ήθελε να επιβάλλει στον Καναδά για συγκεκριμένα καύσιμα. Ε, η αντίστοιχη είναι η κατάσταση και με τον Καναδά ε, και στο κεφάλαιο της βιωσίμου ανάπτυξης. Και εδώ κινδυνεύουμε είτε να αποδυναμώσουμε το σχέδιο της αντιμετώπισης της αποψήλωσης των δασών ή των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, διακινδυνεύοντας αυτά που προσπαθούμε να πετύχουμε και διακινδυνεύοντας και τις δυνατότητες του να βελτιώσουμε κάτι που δεν έχουμε ακόμα ψηφίσει. Όχι μόνο τι θα μπορούσαμε να πετύχουμε σήμερα δηλαδή και να γίνει αυτό σεβαστό, αλλά αυτά που πιο αργά θα χρειαστεί να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το φινικέλαιο και το θέμα αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί εν ώψη του 2030. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Διότι η αγορά των αγροκαυσίμων είχε, είχε πραγματικά εντυπωσιακά αυξηθεί αλλά υπάρχουν σημαντικότατες ανησυχίες σχετικά με τις εκπομπές θερμοκηπίου. Τώρα, πέραν αυτού υπάρχει το θέμα των ε, διαιτητικών δικαστηρίων, ε, των ε, μηχανισμών επίλυσης διαφορών, ISDS e και τα λοιπά. ISDS. E Η Ινδονησία μέχρι τώρα αντιστεκόταν ε, σε αυτό το θέμα και μάλιστα δεν έχω καταλάβει ακριβώς πού βρισκόμαστε με την Ινδονησία ως προς αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα βασικότερα θέματα ε, δηλαδή για το φινικέλεο δεν μπορώ να φανταστώ ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι η Κομισιόν θα ήταν τόσο σχιζοφρενική ώστε να θέλει να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον, το κλίμα κτλ. και τους βατράχους αφενός και αφετέρου να θέλει να προστατεύσει και τα οικονομικά συμφέροντα επιχειρήσεων που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μινόχ για την ΚΟΕ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόεδρε, υπογράφει συμφωνίες ε, με διάφορες χώρες στον κόσμο. Αναρωτιέμαι όμως τι σημαίνει αυτό για τους δικούς μας πολίτες, αλλά και για τους πολίτες Ινδονησίας. Έχουμε το θέμα της αποψήλωσης των δασών και των ελαίων και των φαρμάκων. Το φινικέλαιο θα έπρεπε να αποκλείεται τελείως από τη συνθήκη αυτή γιατί είναι επικερδές για τους 14 εκ των ε, πολυδισεκατομμυριούχων στην Ινδονησία και απολύτως καταστροφικό για όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Έχει σχέση με την εγκληματικότητα, έχει σχέση με τις πυρκαγιές τις στιμένες πυρκαγιές, την καταστροφή των δασών, την, τον εκδιωγμό ανθρώπων από τα σπίτια τους, η οδηγία θα έπρεπε να εξαιρεί το φινικέλαιο. Πρέπει να είμαστε πιο ρητοί εμείς. Η καταστροφή των δασών είναι κίνδυνος όχι μόνο για τον τοπικό πληθυσμό, για τους πολίτες της αλλά για όλους τους πολίτες του κόσμου μέσω των εκπομπών και η καύση των δασών ε, δημιουργεί προβλήματα με το διοξίδιο, δημιουργεί και προβλήματα δημόσιας υγείας όπου μας οδηγεί και στο θέμα των φαρμάκων. Φαρμακευτικών προϊόντων που δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και προβλέπουμε προεκτάσεις διπλωμάτων, ισχύω διπλωμάτων δηλαδή για συγκεκριμένα σκευάσματα, και το οποίο μας οδηγεί και στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί υπάρχει και το, και το ε, θεμελίως δικαίωμα της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έχω λοιπόν εντονότητα τις αμφιβολίες για τις συμφωνίες αυτές. Είναι καλές για τις πολυεθνικές και πολύ κακές για τους ανθρώπους. Είναι, είναι τέτοιο παραδείγμα. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Χάουταλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο και περίπλοκο το θέμα του φινικέλεου. Έχουμε σημειώσει ότι η Ινδονησία και η Μαλαισία είναι η, η μεγαλύτερη παραγωγή και υπήρξαν εξαιρετικά ενεργές τους τελευταίους μήνες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ είχα επαφές με, μαζί τους, με τους εκπροσώπους τους και την περασμένη εβδομάδα στην εντολή, μάλλον στο πλαίσιο της συζήτησης ε, των Υπουργών ΑΣΕΜ, είχε συσταθεί μια ομάδα εργασίας μεταξύ της ΑΣΕΑΝ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους παραγωγούς φινικελαίου. Αυτή η ομάδα εργασίας τι θα μπορούσε να επιτύχει και πώς συνδέεται αυτή η δουλειά με την προθεσμία δημοσίευσης κομισιών της κατεξιοδότησης πράξης για την οδηγία ανανεωσίμων. Η καλύτερη προσέγγιση που θα μπορούσαμε να έχουμε θα ήταν μια διαφάνεια στην αλυσία προμήθειας. Λογοδοσία δηλαδή στην αλυσία προμήθειας. Και η φλεγ της Ινδονησίας ακριβώς σε αυτό στοχεύει στην νομιμότητα των προϊόντων ξυλία μεταξύ άλλων. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια προσέγγιση λογοδοσίας της ε, ε, αλυσίδα προμήθειας αντίστοιχη με αυτά που κάνουμε για τα προϊόντα δασοκομεία. Η κατεξιότητα πράξη, λένε αρκετοί συναδελφοί, είναι κρίσιμη σημασία για να βρεθεί βιώσιμη λύση στο πρόβλημα αυτό. Ό,τι μηχανισμό και να έχουμε τελικώς. Ε, το σχέδιο δράσης για την αποψήλωση και καταστροφή των δασών που ε, ε, επιτέλους εκκίνησε η Κομισιόν έχει, ενέχει κάποιες διαστάσεις πιο μακαροπρόθεσμης λύσης καθότι έχω επισκεφθεί και τις δύο χώρες αυτές πρέπει να πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι δεν είναι ακριβές ότι δημιουργεί πλότο μόνο για τους δισεκατομμυριούχους, το φινικέλαιο και μιζέρια και καταστροφή για τους υπόλοιπους. Ε, ε, ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες έχουν βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής τους μέσω της οικονομίας που βασίζεται στο φινικέλαιο. Και οι χρήστες του προϊόντος αυτού στην Ευρώπη ε, λένε, πιστεύουν ότι οι μικρομεσαίοι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να συμμετάσχουν στο σύστημα. Είναι λοιπόν δύσκολο το θέμα. Δεν μπορούμε απλά να πούμε ας πάψουμε να εισαγάγουμε και εδώ να πούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένοχη. Γιατί έχουμε τον κανονισμό για το μείγμα ανανεωσίμων στα βιοντίζελ. Υπήρξαμε υπερβολικά ενθουσιώδης για τα αγροκαύσιμα. Και ίσως η αγορά δείχνει ότι δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα πέρα από όλες τις υπόλοιπες ανησυχίες και επομένως και ως καταναλωτές έχουμε ευθύνη να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Κύριε. Κιόνιχ. Σας ευχαριστώ για πολλές και καλές ερωτήσεις γνωρίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται στην παρούσα φάση για το RED 2 την κατεξουσιοδότηση πράξη. Όπως είπε ο εισηγητής, οι σχέσεις με την Ινδονησία μέχρι τώρα έχουν τεκμηριώσει το θέμα της συμβατότητας της ε, πρότασης αυτής. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική κατάληξη, αλλά παρακολουθούμε ε, με προσοχή το τι συμβαίνει σε σχέση με την ε, κατεξουσιοδότηση πράξη. για τις επιφυλάξεις για το φινικέλαιο και τις επιπτώσεις στο φτωχό πληθυσμό είναι βασικό προϊόν στην Ινδονησία στα πλαίσια της καταπολέμησης της φτώχειας και της αύξησης των θέσεων εργασίας. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο η ίδια η Ινδονησιακή κυβέρνηση ε, προσπαθεί να εμπλέξει όσο μπορεί περισσότερο ε, τα στενέστερα τμήματα της κοινωνίας έτσι ώστε οι καλλιέργειες φινικελαίου να είναι ε, βιώσιμες. Δεν έχει ολοκληρωθεί φυσικά αυτή η διαδικασία, αλλά έχουμε κάθε συμφέρον να προχωρήσουμε σε διάλογο με τους Ινδονήσιους μέσα από προγράμματα τα οποία θα διασφαλίσουν την ισορροπία ανάμεσα στο βιώσιμο κομμάτι ε, της καλλιέργειας, τους στόχους της χιλιετίας, και τον θεμητό επίσης στόχο καταπολέμησης της φτώχειας και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Υπάρχει επίσης και το θέμα της αύξησης της απόδοσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Τα θέματα όλα αυτά όμως ε, είναι υπό εξέταση ακόμα και σε επίπεδο σχεδιασμού και φυσικά σε επίπεδο εφαρμογής εμείς και σε εσωτερικό νομικό επίπεδο μέσω των οδηγιών και σε σχέση με τον κανονισμό για τα δάση τα που έχει ήδη προταθεί και είναι υποδιαβούλευση να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι αιτίες επί της ουσίας και τα αρνητικά αποτελέσματα. Είναι βασικό προϊόν για την Ινδονησία, είναι το 50% των εξαγωγών της επίσης και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε το σύνολο των προϊόντων και των αγαθών γενικότερα, τα οποία είναι αντικείμενα εμπορίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά η εξαίρεση του φινικελαίου δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από πλευράς μας. Είναι αλήθεια ότι άνω των 60 εκατομμυρίων ε, μικρών ιδιοκτητών ή μικροϊδιοκτητών εμπλέκονται και φύγονται από πιθανές ρυθμίσεις στον τομέα του φινικελαίου. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εισαγωγές δεν είναι παρά το 12% στην Ένωση ενώ της παραγωγής της Ινδονησίας. Οπότε ακόμα και αν λάβουμε μέτρα δεν πρόκειται να λύσουμε εμείς το σύνολο του θέματος. Παρ' όλα αυτά απαιτείται περισσότερη εμπλοκή και συμμετοχή και των υπόλοιπων εταίρων. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες χώρες οι οποίες εμπλέκονται περισσότερο από εμά. Σε σχέση με όλα αυτά να πω επίσης και για την ομάδα εργασίας του ΑΣΕΑΝ για το Φινικέλαιο. Ε, υπήρξαν κάποια στοιχεία ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε που θα καταλήξει ο διάλογος, αλλά είναι επίσης σαφές ότι απαιτείται περισσότερος διάλογος, θα γνωρίζουμε έτσι το πού βρίσκεται η κάθε χώρα, τι πιστεύει η κάθε χώρα και έτσι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε καλύτερα χώρες όπως η Ινδονησία αφού λάβουμε υπόψη φυσικά τις βασικές αιτίες του προβλήματος. Ένα άλλο θέμα είναι ότι το 50% ε, του ε, φινικελαίου που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γίνεται χωρίς επιβολή δασμών, όχι το σύνολο. Παρ' όλα αυτά επαναλαμβάνω το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι τα κριτήρια μέσα από τα οποία γίνεται η εμπορία του φινικελαίου. Και φυσικά υπάρχουν και από πλευρά της βιομηχανίας αρκετές σκέψεις στην παρούσα φάση που θα οδηγήσει τη βιομηχανία να συμμετέχει και να ενδιαφέρεται για τις συζητήσεις αυτές. Για τη σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ε, πράγματι, ε, το θέμα της ε, έχουν μεν επικυρώσει, αλλά το θέμα της εφαρμογής είναι το πρόβλημα και το θέμα της εποπτείας επίσης και του αναφέρεστε σε σχέση με την εφαρμογή. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων στον τομέα αυτό είναι ε, σαφής. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούν και επιδιώκουν να πετύχουν οι Ινδονήσοι και γι' αυτό ακριβώς επικυρώνουν όλες αυτές τις συμβάσεις. Τώρα για τα δικαστήρια τα διαιτητικά είναι τμήμα της διαπραγματευτικής εντολής, είναι τμήμα της διαπραγμάτευσης μέχρι τώρα. Προ στιγμήν οι Ινδονήσοι δεν έχουν πει ότι είναι έτοιμοι να ε, προσυπογράψουν. Βλέπουμε σε ποια φάση βρίσκονται οι ενδιάμεσες διαπραγματεύσεις. Όπως γνωρίζετε οι Ινδονήσοι πήραν την απόφαση να τερματίσουν τις δικές τους διμερείς ε, δικαστικές ε, φόρμουλες σε ε, για μια χώρα σαν την Ινδονησία θα πρέπει να υπάρξει κάτι για τους ε, επενδυτές γιατί δεν έχουν θα έλεγα το λεγόμενο τέλειο ε, σύστημα ρύθμισης που προβλέπεται για το συγκεκριμένο θέμα από ένα κράτος δικαίου αλλά όλα αυτά είναι ανοιχτά προς διαπραγμάτευση. Τώρα για τις περιοχές, τις φυσικές περιοχές που ανήκουν στις οδηγίες Habitat ε, και τα, την πανίδα που απειλείται ε, σύμφωνα με τα θέματα τα οποία επιβάλλει προς εξέταση η σύμβαση ΣΑΙΤΕΣ. Το θέμα έχει έρθει στην ημερήσια διάταξη, συμπεριλάβαμε το θέμα αυτό, θα πρέπει να δούμε πώς το θέμα αυτό θα συμπεριληφθεί στα ισχύοντα προγράμματα και είναι κάτι βέβαια για το οποίο και οι ίδιοι Ινδονήσοι ανησυχούν. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσεις ακριβώς γιατί θα είναι τμήμα των ε, συζητήσεών μας από εδώ και πέρα. και όταν κυκλοφορήσει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο η ενδιάμεση έκθεση θα έχουμε την άνοιξη άλλωστε και την έκθεση του Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο. Τώρα για την πρόσβαση στα φάρμακα. Δεν θα υπάρξει κάτι στη συμφωνία το οποίο θα μπορούσε να εμποδίσει τους ε, Ινδονήσιους να παράγουν statement on, on... Τα γενώσιμα φάρμακα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, υπάρχουν προβλέψεις οι οποίες το επιτρέπουν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους Ινδονήσιους ε, να διαθέτουν φάρμακα στους πολίτες τους ε, σε λογικές τιμές. Το θέμα λοιπόν, όπως και στις υπόλοιπες μορφές διαπραγμάτευσης, είναι να υπάρξει μια σωστή ισορροπία ανάμεσα τα δικαιώματα τα οποία έχουν ε, οι πολίτες για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν ε, ή μάλλον για να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες σε λογικές τιμές. Η συμφωνία αυτή πάντως δεν περιλαμβάνει κάτι το οποίο θα δυσκολέψει τους Ινδονήσιους στην παραγωγή γενοσύμων. Καλώς σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κένιχ. Νομίζω ότι είναι μια ιστορία η οποία θα κρατήσει αρκετά. Σας ευχαριστώ, θα μείνουμε σε επαφή. the last, item for today is the... Το τελευταίο θέμα για σήμερα είναι το 31. Ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στον τομέα των ελευθέρων συμφωνιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη της έκθεση εδώ και λίγες εβδομάδες. Συζητήσαμε σε βάθος την πρώτη έκθεση και είχαμε πει ότι θα θέλαμε να υπάρχουν πιο ξεκάθαρες ε, αναφορές στις επιπτώσεις ε, για τους τοπικούς πληθυσμούς. Διευκρινίσαμε επίσης ότι θα πρέπει να δούμε το τι ακριβώς γίνεται με την ε, χρήση των, των συμφωνιών ε, προτιμησιακών σχέσεων για συγκεκριμένα προϊόντα και συγκεκριμένες χώρες. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κάνει την παρουσίασή της για 8 λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ με μεγάλη χαρά. Θα σας μεταφέρω αυτά τα οποία έχουμε ολοκληρώσει στην δεύτερη ενδιάμεση παρουσίαση. 35 συμφωνίες με 62 εταίρους. Έχουμε και κάποια τεχνικά στοιχεία τα οποία μπορούν να σας δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε χώρα και για κάθε συμφωνία. Να σας πω ότι η έκθεση διευθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες στόχους. Λοιπόν, έχουν λειτουργήσει, έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις των οικονομιών τις οποίες καλύπτουν αυτές τις συμφωνίες και φυσικά έχουν προωθήσει τις ευρωπαϊκές αξίες και έχουν υποστηρίξει τις υπόλοιπες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την πολιτική για την ανάπτυξη. Επί τη βάση αυτών των τριών στόχων τα FTA συνεχίζουν να βοηθούν στο άνοιγμα των αγορών, στην αύξηση των εξαγωγών. Το είδαμε αυτό ε, με την αύξηση κατά 10% ε, η οποία σημειώθηκε μέσα από την υπογραφή των συμφωνιών δεύτερης γενεάς και όπως είπατε έχουμε ε, ε, χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες κατά προτίμηση εξαγωγών από τις χώρες αυτές ε, κατά 80 περίπου της 100, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Έχουν ε, υπάρξει επίσης προσπάθειες για απόσυρση εμποδίων, ιδιαίτερα στον τρομέα των τροφίμων Έχουμε προχωρήσει στην καταγραφή φαρμακευτικών και χημικών ουσιών σε χώρες όπως το Μεξικό και έχουμε ε, διευκρινίσει κάπως τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν σε σχέση με την Ουκρανία και την Τουρκία. Είπα ότι έχει υπάρξει βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου. Ε, υπήρξαν κάποια βήματα για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, όπως είπα, η Ουκρανία υιοθέτησε ένα οδικό χάρτη για τις δημόσιες προμήθειες και το Μεξικό απέσυρε κάποια από τα εμπόδια τα οποία υπήρχαν για την εφαρμογή της συμφωνίας. Τώρα για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών έχει υπάρξει ε, πρόοδος και στον τομέα ε, των ε, εργασιακών δικαιωμάτων και στα πλαίσια της ε, σύνθεσης ε, των ε, συμβουλευτικών ομάδων γύρω από τη λειτουργία της ΣΕΤΑ. Ε, υιοθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο ε, τρεις συστάσεις και για τον τομέα του σεβασμού των αποφάσεων για τη μετρία των συνεπειών για τις κλιματικές αλλαγές. Έχουμε λοιπόν να πούμε ότι συνολικά σε σχέση με τις εξαγωγές από τις χώρες αυτές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 10 χρόνια σημειωθεί αυξήσεις που φτάνουν το 70%. Ε, θα επανέλθω και στις συστάσεις τις οποίες μας έστειλε το Κοινοβούλιο το Μάιο του 2018 ε, κανόνες για ε, την αναφορά της προέλευσης των προϊόντων, τομεακές αναλύσεις ε, του αγροτροφημικού τομέα και επίσης βελτίωση των εταιρικών σχέσεων ε, και επίσης βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στα όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη. Τώρα μιλήσαμε για τα καλά σημεία, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και δυσκολίες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, αναφερθήκατε κι εσείς στην εισαγωγή σας, εμείς ε, παρόλες τις εξελίξεις τις θετικές υπάρχουν ε, όμως πολύ περισσότερες δυνατότητες και αν χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες αυτές ε, η ε, δυνατότητες, ε, υπάρχει δυνατότητα εξοικονόμησης σε επίπεδο δασμών που ξεπερνάει τα τρία δις ε, για τον επόμενο χρόνο. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την χρήση των συμφωνιών, κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Η δεύτερη κατηγορία των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε είναι τα μη δασμολογικά εμπόδια, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου. Υπάρχει το θέμα, ας πούμε, προστατευτικών μέτρων στα πλαίσια των διαδικασιών πιστοποίησης για κάποια κυκλοφορία νέων προϊόντων. Υπάρχει επίσης και έλλειψη διαφάνειας. Αν μία επιχείρηση δεν γνωρίζει ακριβώς τους κανόνες για τους δημόσιους διαγωνισμούς και τις προμήθειες, κρατικές προμήθειες, τότε είναι προφανές ότι ε, φύγεται η ανταγωνιστικότητά της. Ε, θα τελειώσω τώρα με τρεις ε, γενικότερες σκέψεις. Καταρχά θα φύγω λίγο από τα στατιστικά. Καταρχάς βρισκόμαστε πάντα σε μια διαδικασία μαθητείας Έχουμε ξεκινήσει να επεξεργαζόμαστε τώρα την τρίτη έκδοση της συγκεκριμένης έκθεσης. Έχουν δημιουργηθεί πραγματικά πάρα πολλές επαφές ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και τις υπόλοιπες Γενικές Διευθύνσεις, όπως επίσης και το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Εμείς λοιπόν διαπραγματευόμαστε και αυτό είναι καλό όχι μόνο για την Επιτροπή αλλά για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες της Ένωσης. Όταν βλέπουμε τους αριθμούς διαπιστώνουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να υπερεκτιμήσει κανείς τη σημασία των FTAs. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν λειτουργούμε εν κενό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία παίζουν ρόλο όπως οι μακροοικονομικές εξελίξεις, οι γεωστρατηγικές εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο και ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλοι εταίροι οικονομικοί με τους οποίους ε, οι χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε προχωρούν σε ε, συμφωνίες. Πάντως, οι συμφωνίες αυτές δημιουργούν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αν θέλετε, αντιμετώπισης των προβλημάτων γύρω από τα θέματα συμμόρφωσης με τους όρους της συμφωνίας. Ε, μπορούμε επίσης σε τεχνικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο να παίρνουμε ένα βήμα επιπλέον, όχι μόνο σε επικοινωνία με τα Υπουργεία Εμπορίου, αλλά και ε, πάνω από αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Οι επιτροπές αυτές λοιπόν δεν έχουν μόνο σαν στόχο να φέρνουν στην επικαιρότητα τα θέματα συμμόρφωσης και σεβασμού, αλλά γενικότερα θέματα κοινού συμφέροντος όπως διαφορετικές μορφές συνεργασίας. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η ΣΕΤΑ. Εμείς είχαμε συζητήσει και εξακολουθούμε να συζητούμε με τους Καναδούς το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε από κοινού βήματα πρόοδου στον τομέα του κλίματος. Ε, δεν είναι μόνο αριθμοί και στατιστικές οι συμφωνίες αυτές. Αν και κατανοώ βέβαια ότι αυτά τα οποία διαβάζετε στην έκθεση είναι ένα αισθαντανέ αυτού που έγινε το 17. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μια γενικότερη ακόμα. Συγγνώμη μακρηγόρησα. Ευχαριστούμε λίγο πρόεδρος. Παρακαλώ συνάδελφε, θέλετε να παρέμβετε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το θέμα είναι τι κάνουμε με τις εκθέσεις που εδώ συντάσσουμε, παράγουμε. Αν υπάρχουν κάποια στοιχεία στα οποία επιθυμούσε να συνεισφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο ΣΕΤΑ, ήταν τα κλιματικά, τα περιβαλλοντικά. Συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων και όχι μόνο εκθέσεων. Ο Καναδάς, παρά τον ενθουσιασμό που εκφράζει ο Πρωθυπουργό του κάποιες φορές δεν έχει καθόλου ενεργειακή πολιτική συμβατή προς την προστασία του περιβάλλοντος. Και μάλιστα εμείς έχουμε αυξήσει τις εισαγωγές καυσίμου. Ορυκτών καυσίμων δηλαδή. Και ε, και σχιστολιθικού. Η εντύπωσή μας λοιπόν είναι ότι στο βαθμό που οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, είναι σε θέση να κινηθούν ώστε νομικά να, είναι, να, συμμορφού, να συμμορφούνται, τόσο οι μικρότερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται ε, να προσαρμοστούν διότι προτιμούν αντί να αναλάβουν ένα τέτοιο υψηλό άχθος ε, προσαρμογής να πληρώσουν ένα μικρό πρόστιμο. Ο πρόεδρος. Εγώ πρόσφατα στην τηλεόραση άκουσα μια, παρακολούθησα μια συνέντευξη με αντικείμενο την Γκάνα. Η εξαγωγή λοιπόν κακάο λόγω της IPA αυξάνεται αλλά η κατάσταση των ανθρώπων στην Κάνα δεν έχει βελτιωθεί λόγω των αυξημένων αυτών εξαγωγών και οι Γκανέζοι φεύγουν από τη χώρα πάνε στην Ιταλία, δουλεύουν στην καλλιέργεια ντομάτας η οποία μετά εξάγεται στην Κάνα. Ντομάτα. Και μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται υπό πολύ σκληρές συνθήκες στην Ιταλία, άδικες. Επομένως, η IPA ήταν προς το συμφέρον των Γκανέζων. Αυτή είναι η ερώτηση δική μου, λέει ο πρόεδρος. Πολύ καλή ερώτηση, Πρόεδρε. Πολύ καλή ερώτηση. Πέρσι τον Οκτώβριο είχαμε μια μελέτη για την καλή ισορροπία μεταξύ τέλος πάντων πλέον εκτιμάτων και μειονεκτιμάτων των FTA. και από τα πορίσματα προκύπτει ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ακόμα και μεσοπρόθεσμη βελτίωση στις χώρες εταίρους όσο στη δική μας οικονομία. δεδομένης της ανησυχίας που εκφράζεται από την πλειοψηφία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε κατανοήσει τον πλήρη αντίκτυπο των κοινωνικό, κοινο, οικονομικό και περιβαλλοντικό των πολιτικών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μήπως βλέπουμε τις FTA ως μέσο ανταγωνισμού εξαγωγής μάλλον του ανταγωνισμού από την εσωτερική μας αγορά σε τρίτες χώρες. Έχουμε λάβει μακροπρόθεσμα υπόψη μας το συμφέρον των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των πολιτών ή απλώς συνεχίζουμε με την έννοια του ανταγωνισμού εξάγοντας την από εσωτερική αγορά σε τρίτες χώρες οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικούς παράγοντες από τους δικούς μας και με υποδιαφορετικά οικονομικά μοντέλα. Είναι πράγματι η FTA το εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει να επανεξετάσουμε το δικό μας οικονομικό-κοινωνικό μοντέλο πρότυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι μόλις χθε είχαμε μια ανακοίνωση τύπου ότι ακριβώς όπως είπατε και εσείς ο Καναδάς καθόλου δεν σέβεται τις περιβαλλοντικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρωτόκολλο. Και πολύ συχνά σήμερα όπως κάθε πέμπτη έχουμε διαδηλώσεις εδώ στο Βέλγιο. Κλιματικές. Και αν δεν δούμε το πώς και οι FTA συνεισφέρουν σε αυτό το πρόβλημα, τότε δεν τηρούμε και τις υποχρεώσεις μας προς τους εταίρους μας. Μεγάλα ερωτήματα τα οποία δεν είναι τόσο εύκολο να απαντηθούν, αλλά έχουμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Παρακαλώ λοιπόν. Νομίζω πως ε, το πρώτο ερώτημα αφορούσε τη ΣΕΤΑ και το κεφάλαιο και ε, το ερώτημα του γιατί δεν κινούμαστε απευθείας προς τον μηχανισμό επιπολής κυρώσεων. Όπως γνωρίζετε ξεκινήσαμε ε, αυτό το, την, την, την χάραξη αν θέλετε του σχεδίου δράσης των 15 σημείων όπου περιλαμβάνουμε όλους τους stakeholders, όλα τα σημεία που θα πρέπει να εφαρμοστούν, ε, και ξεκινούμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία στο πλαίσιο όλων των 7 συμφωνιών ε, Κολομβία, Περού, Καναδάς και το καθεξής και στις επιτροπές ε, και στην κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να προωθήσουμε ακριβώς την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Και σας λέω ότι εξετάζουμε αυτή την περίοδο τις προτεραιότητες της εκάστοτε χώρας πολύ συγκεκριμένα, το κάνουμε δηλαδή με τους εταίρους FTA και από εκεί και μετά εάν ε, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό ε, το σχέδιο δράση δεν λειτουργεί καλά, έχουμε προβλέψει για ένα μηχανισμό αναθεώρησης. Πάντω, σε γενικέ γραμμές, η θέση της Επιτροπής ήταν ότι δεν ε, δεν αποφέρει περισσότερα αποτελέσματα ο μηχανισμό τη επιβολή ε, σε σύγκριση με αυτό που έχουμε εμεί προβλέψει με βαστή ΣΕΤΑ. Ε, και ε, κυρίω ε, οι μεγάλε επιχειρήσει είναι εκείνε που υποφελούνται από τι FTAs. Και ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν ε, έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Υπάρχει έλλειψη δεδομένων ω προ το κατά πόσο οι εξαγωγέ από πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποφελούνται και αξιοποιούν δηλαδή τις ευθείες. Πάντως ε, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτή την πτυχή και μπορώ να σας ενημερώσω πως όλα μας τα project που αφορούν στην, ε, ε, ε την, και τη βάση δεδομένων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εστιάζουν στις ειδικές στι πολύ συγκεκριμένε ανάγκε των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό που κάνουμε εδώ είναι να εξετάσουμε ε, το πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τι πληροφορίε και σε ό,τι αφορά την παρουσίασή του, αλλά και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του. Δηλαδή, τι ε, καθιστούμε διαδραστικέ, τι ε, διαθέτουμε σε διαφορετικέ γλώσσε, έτσι ώστε οι επιχειρήσει να γνωρίζουν, να καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν ακόμα πού μπορούν να λάβουν περισσότερε πληροφορίε, δηλαδή ε, σύνδεσμοι στο σύνδεσμο άλλων γενικών διευθύνσεων και ούτω καθεξής. Και επίσης προβλέπουμε πως φέρουμε και σεμινάρια. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με την Ιαπωνία έχουμε ξεκινήσει κάποια webinars ε, και στο πλαίσιο της ΣΕΤΑ επίσης. Ε, ερχόμαστε σε επαφή και μέσω των κρατών μελών, για παράδειγμα με οργανώσεις επιβιώσουν, ώστε ακριβώς να υπάρχει μια καλύτερη αντίληψη του ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τι χρειάζονται. Ε, και επίσης λαμβάνουμε υπόψη μας και το έγγραφο που κατάρτισε το Eurochamber σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράση. Μετά, σε ό,τι αφορά τα έτες και ε, το παράδειγμα της Γκάνα που αναφέρατε, ναι, οι αξαγωγέ αυξήθηκαν και συγκεκριμένα στο Καμερούν σε ό,τι αφορά τα προϊόντα κακάο και συχνά ακούμε ότι οι τοπικοί παραγωγοί δεν επωφελούνται όσο θα έπρεπε ή αντιθέτως ε, υποβάλλονται ε, σε, σε, ε, σε αρνητικό αντίκτυπο ε, με βάση αυτές τις συμφωνίες, αλλά με βάση τους εμπειρογνώμονες συναδέλφους μου από τους 29 εταίρους στις IBS δεν έχουμε διαπιστώσει δραματική αύξηση των εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν ναι, κάποιες περιπτώσεις όπου η κατατόπους ε, ε, παραγωγή δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτή την αύξηση των εξαγωγών από την πλευρά τους. Και όπως γνωρίζετε έχουμε και την υποστήριξη που προφέρουμε για παράδειγμα 6 δισεκατομμύρια από το 2016 αλλά και μέσω του νέου μηχανισμού του σχεδίου σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Και Προσπαθούμε τώρα να δούμε από κοινού με τους συναδέλφους ε, πώς ε, μπορεί αυτός ο μηχανισμός, αυτό το εργαλείο να αποφέρει περισσότερους καρπούς, εξετάζοντας δηλαδή και ειδικότερα τον τρίτο ε, πυλώνα της Συμφωνίας ΕΠΗ. Πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ζήτημα με το οποίο θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε σε μία από τις ε, περαιτέρω εκθέσεις μας. Σε ό,τι αφορά το κατά πόσο FTS αποτελούν πραγματικά ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βελτιώσει ε, την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και το ερώτημα που τέθηκε ως προς το ότι ενδεχομένως να είναι αντιφατικός αυτός ο στόχος σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες. Να σας πω ότι εγώ δεν θεωρώ πως είναι αντιφατικά τα αυτά τα δύο στοιχεία. Δηλαδή πάντοτε θα είμαστε σε ανταγωνισμό με τους ε, εταίρους μας στον πλαίσιο των συμφωνών FTA. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τα πράγματα έτσι ώστε η ανταλλαγή, η κυκλοφορία, η, αγαθών και υπηρεσιών να διευκολύνεται. Και νομίζω πω ε, μπορούν να βελτιωθούν πολύ περαιτέρω τα πράγματα και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, του ίσους όρου του παιχνιδιού. Και το αναφέρομαι ειδικότερα στα ε, δικαιώματα ε, διανοητική ιδιοκτησία, σε ό,τι αφορά του κανόνε, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, του περιβαλλοντικού κανόνε. Άρα λοιπόν πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα για να βελτιώσουμε ακριβώ του, το, τους ίσους όρους του παιχνιδιού. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ζήτημα εδώ των δασμών που μας αφορά, γιατί πράγματι όπως έχετε πει ε, βλέπουμε συχνά κάποιες επιχειρήσεις να μην αξιοποιούν ε, τις ε, συμφωνίες FTA γιατί είναι υπερβολικό το γραφειοκρατικό άκτος. Δηλαδή αν οι δασμοί για παράδειγμα στο πλαίσιο μιας ε, σε σχέση με μια χώρα είναι σχετικά χαμηλή, προτιμούν να υποβάλλονται στους δασμούς. Αλλά σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τους κανόνες ε, ε, προέλευσης και πολλά άλλα ζητήματα, ότι να κάνουμε τα πάντα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διευκολύνουμε την αξιοποίηση των συμφωνιών FTA. Δεν θα πρέπει δηλαδή να επαναπαυόμαστε. Έχουμε επιτύχει καλά αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα και χρειαζόμαστε επίση καλύτερα περισσότερα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ε, στο πλαίσιο για παράδειγμα της ΕΤΑ είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί για παράδειγμα το 35% των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Καναδά είναι υπηρεσίες οπότε θα πρέπει να έχουμε περισσότερα δεδομένα ούτως ώστε να γνωρίζουμε το πώς επηρεάζει αυτή η αυξημένη παροχή υπηρεσιών ε, τους ανταγωνιστές μας και εμάς. Άρα λοιπόν αυτά προσπαθούμε να επιτύχουμε αποκινούμε εσά και με του εμπειρογνώμονέ μα, ούτω ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια συμπληρωματική ερώτηση από τον κύριο Σόλτς. You are not the right addresser for, for this debate, maybe alone. Ίσως δεν ε, θα πρέπει να θέτω σε εσά το ερώτημα αυτό. Ποια είναι η διαδικασία στο εσωτερικό της Επιτροπής ε, για τα συμπεράσματα της έκθεσής σας που είναι ενδιαφέροντα, αλλά πώς εσείς οργανώνετε την επικοινωνία των απόψεων με τις υπόλοιπες γενικές ε, διευθύνσεις σχετικά με την εφαρμογή των ε, ε, συστάσεών σας, των συμπερασμάτων σας. Γίνεται μια κάποια συζήτηση για να γνωρίζουν αυτά τα οποία κάνετε. Λοιπόν, σαφής η ερώτηση, παρακαλώ μια σαφή απάντηση. Οι υπόλοιπες γενικές διευθύνσεις έχουν ε, ήδη ε, συζητήσει και διαβουλευτεί τα θέματα αυτά στο εσωτερικό, για τα θέματα αυτά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργάζομαι και με τους υπόλοιπους συναδέλφους, ε, με τις άλλες γενικές διευθύνσεις σε συγκεκριμένα θέματα για θέματα ας πούμε προστασίας των δασών, για θέματα ε, φορολογίας. Ε, γενικά υπάρχουν γενικές διευθύνσεις που έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και γι' αυτά συζητάμε τώρα. Υπάρχει επίσης η έκθεση που στείλαμε στους υπουργού της 9 Νοεμβρίου για το εξωτερικό εμπόριο και η Γενική Διεύθυνση έχει δημιουργήσει και μια ανεπίσημη ομάδα εργασίας πέρυσι η οποία συναντιέται δύο-τρεις φορές το χρόνο και όπου οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών για τα θέματα της εφαρμογής των FTA συζητάνε και αναφέρονται στις εξελίξεις, στις νέες μελέτες, στις νέες ε, εξελίξεις και στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Και επίσης έχουμε και τις εκθέσεις εφαρμογής, έχουμε επίσης και την ομάδα εμπειρογνωμόνων για ε, την αηφορία στην ανάπτυξη που συναντιέται τέσσερις φορές το χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω λοιπόν η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί και να οδηγήσει σε κάποια νέα επιμέρους στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά. Κλείνουμε λοιπόν με το 32. Όχι με το 31, το 32 τώρα δεν ξέρω, ε, δεν είναι στα διάφορα. Η επόμενη είναι συνάντησή μας 4 Φεβρουαρίου και μετά 18 και 19 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.